Λοιπόν, τα εγκρίνει τη μερσιά διάταξη. Τα πρακτικά τη περισμένη συνεδρία τα έχετε μπροστά σα. Αν μέχρι το τέλο τη συνεδρία σα δεν έχετε παρατηρήσει, αν μα πείτε κάτι θα το διορθώσουμε. Αλλιώ θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Περνάμε στι ανακοινώσει του Προέδρου, σημείο 3 τη ημερησία διάταξη. Περνάει στο web stream η συνεδρία αυτή, ο συνήθω. Έχουμε διερμηνία και σήμερα και αύριο σε όλες τις γλώσσες εκτός από σφιδικά, εσθονικά, λιδωνικά ε, και μαλτέζικα. Όλες οι άλλες γλώσσες υπάρχουν. σήμερα τέσσερις ημερες διάταξης. Παρουσίαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Έχουμε μια νέα προεδρία στο Συμβούλιο, τη Βελγική. Και έχουμε σήμερα τρεις υπουργούς. Μεγάλη μας τύχη να τους ακούσουμε. Καταρχήν, την Υπουργό Πολιτισμού Οδοκαστικού Τομέα Υγείας και Ισότητας των Ευκαιριών της γαλλόφωνης κοινότητας του Βελγίου. Ελπίζω να μην ξέχασα καμία από τις ε, αρμοδιότητες γιατί είναι δύσκολο το Βέλγιο σε αυτά. Ναι, γιατί είναι ομοσπονδιακή χώρα και γι' αυτό εκπροσωπούνται διάφορες ομάδες. Η Υπουργός κυρία Λάνεν είναι υπεύθυνη για τον πολιτισμό, τα από του και μπορώ να της πω ότι έχουμε κάποιες σημαντικές εκθέσεις που συζητάμε αυτή τη στιγμή με την κυρία Σάντσα Σμιθ που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι ακόμα εδώ το θέμα της ε, πολιτιστικής ε, και δημιουργικής βιομηχανίας μετά ο Ρωσαμίναξης Τρούιπερ για το θέμα Ευρωπαϊκά ε, ολοκλώθηκε η έκθεση, δηλαδή δεν έχει περάσει από το Συμβούλιο και θα πρέπει το Συμβούλιο να προσπαθήσει νομίζω να δώσει στην Ευρωπαϊκή το πρόσωπο του πολιτισμού μας που θέλουμε και γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα, χρειαζόμαστε τότε να βρούμε δωρητές. Αλλά αυτά είναι πράγματα που μπορεί να φροντίσει το ίδιο το Συμβούλιο εκάστοτε για κάθε χώρα. Μετά έχουμε την ανακοίνωση της Κομισιόν για τον κινηματογράφο και την προστασία της οπτικοακουστικής κληρονομιάς. Μετά έχουμε την ε, ε, της κληρονομιάς, ένα θέμα που εξετάζει η κυρία Παλιαρδέλη, που ελπίζω να έρθει. Είχαμε πολύ καυτή συζήτηση του θέματος και γι' αυτό ελπίζω ότι στο τέλος να έχουμε μια κοινή προσέγγιση. Να μην απομονηθούμε δηλαδή πολύ από τις ε, ιδέες της, ε, του Συμβουλίου και μπορεί η κυρία Υπουργό ίσω να μας μεταβιβάσει στο σημείο αυτό την άποψη του Συμβουλίου. Θα ήθελα να προτείνω τώρα να σας δώσουμε τη δυνατότητα σε ένα τέταρτο να μας πείτε κάτι για τον τομέα των αναδοτήτων και μετά μέχρι τις θέσεις θα έχουμε ερωταποκρίσεις και μετά θα ακούσουμε τον επόμενο Υπουργό και ούτως καθεξής. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να υποβάλουν ερωτήσεις μόνο σε θέματα της αρμοδιότητας της Υπουργού. Μετά θα έχουμε τον Υπουργό για το Αθλητικά και για την ε, Νεολαία και την Παιδεία. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, με πολύ μεγάλη χαρά εμφανίζομαι σήμερα μπροστά σας για να ανταλλάξουμε απόψεις για τις προτεραιότητες που θα προωθήσει η Βελγική Προεδρία στη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών. Ο δυναμισμός της Επιτροπής στην οποία συμμετέχετε είναι αναγνωρισμένος και τον εκτιμούν όλοι και είμαι βέβαιη ότι η συνεργασία μας θα είναι επικοδομητική. Θα ήθελα να επιμείνω στο γεγονός ότι και εγώ αλλά και όλη η ομάδα μου που με περιβάλλει στη διάρκεια αυτής της Προεδρίας θα είμαι σε απόλυτη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ανταλλαγή απόψεων στο μέλλον πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Προτού αναφερθώ με πιο συγκεκριμένο τρόπο σε προτεραιότητε τη Βελγικής Προεδρίας, θέλω να σας καθησυχάσω για κάτι. Παρόλο που εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε φάση διαπραγματεύσεων με σκοπό το σχηματισμό μιας νέας ομοσπονδιακή κυβέρνησης, το Βέλγιο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η Βελγική Προεδρία να σταθεί στο ύψο των προσδοκιών που έχετε οι περισσότεροι από εσά για αυτήν. Εξάλλου, ο πολιτισμός και τα οπτικοακουστικά μέσα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κοινοτήτων. Με αποτέλεσμα η επιπτώση των πρόσφατων εκλογών να είναι μηδενικές στη διαχείριση των θεμάτων αυτών από πλευρά μα, Παρόλο που είμαι υπουργό Πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων της κυβέρνησης τη Γαλλική κοινότητα του Βελγίου, το πρόγραμμα που θα έχω την τιμή να σα αναπτύξω σε λίγα λεπτά είναι σαφώς ένα βελγικό πρόγραμμα. Εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφου τη φλαμανδικής και τη γερμανόφωνη κοινότητα οι ε, επαφέ ανάμεσα στις υπηρεσίες και στις διοικήσεις μας, τονίζω επίσης, είναι μόνιμες και θαυμάσιες. Τώρα έρχομαι στι προτεραιότητε τη Βελγική Προεδρία στον τομέα του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων. Αυτέ καθορίστηκαν σε συνεργασία με του ε, εταίρου μα τη τριμερού ομάδα στην Ισπανία και την Ουγγαρία. Ήταν πραγματικά τιμή για μα να είμαστε οι πρώτοι που θα εφαρμόσουμε αυτή τη διάταξη τη συνθήκη τη Λισαβόνα και θα ήθελα να χαιρετήσω την θαυμάσια δουλειά που έγινε από την Αγχέλες Γκονζάλε Σίντε, την Ισπανίδα συνάδελφό μου, τους τελευταίους έξι μήνες. Είμαι βέβαιος ότι έχουμε, βέβαιο ότι έχουμε πραγματικά θέση ορόσημα για το μέλλον. Στον τομέα του πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, θα προωθήσει η Βελγική Προεδρία τέσσερις προτεραιότητες. Πρώτον, θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προβάλλει τις δυνατότητες του κλάδου του πολιτισμού και τη δημιουργικότητας και τους δεσμούς μεταξύ πολιτισμού και καινοτομίας κλάδι, ο πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο έχει αναγνωριστεί σε ουσιαστικό στοιχείο τη καινοτομία και η Προεδρία έχει θέσει σαν στόχο να προχωρήσει προ τη δημιουργία ενό περιβάλλοντο, στο οποίο οι βιομηχανίες αυτές, οι κλάδοι αυτοί θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τι δυνατότητέ του. Όπω προσδιορίζει η Λευκή Βίβλος, ελευθερώνοντα τι δυνατότητε ε, των κλάδων του πολιτισμού και τη δημιουργικότητα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2010 είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε την επιστήριξη που παρέχεται σε αυτό το συγκεκριμένο συγκεκριμένο τομέα προωθώντας τον πολιτισμό σαν πραγματικό καταλήτη της δημιουργικότητας. Αφενός θα καλούμαστε να αποδείξουμε ότι η καινοτομία παίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τομέα και αντιστρόφως ότι ο πολιτισμός αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την καινοτομία στα πλαίσια μιας προοπτικής τόσο οικονομικής όσο και κοινωνικής. Εξάλλου και με βάση αυτή τη διαπίστωση οι εργασίες που θα αναλάβουμε θα έχουν ως στόχο να ανοίξουν νέους οδούς, νέους δρόμους για την ανάπτυξη των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Η ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ανεξάρτητους, στις μικροεπιχειρήσεις και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι οι θεματοφύλακες της πολιτιστικής διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ε, του κλάδου του πολιτισμού και της δημιουργικότητας συμπόσιο θα οργανωθεί για το θέμα αυτό στις Βρυξέλλες 8 και 9 Σεπτεμβρίου, στο οποίο και σας προσκαλώ με ιδιαίτερη χαρά και θα η συζήτηση για τη σχέση μεταξύ δημιουργικότητα πολιτισμού και καινοτομία θα συνεχιστεί εξάλλου στην άτυπη συνάντηση Υπουργών Πολιτισμού που θα λάβει η χώρα στις Βρυξέλλες στις 7 Οκτωβρίου. Δεύτερη προτεραιότητα της Βελγικής Προεδρίας Ο ρόλος του πολιτισμού για την καταπολέμηση τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το έτος 2010 ανακηρύχθηκε ως Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Γι' αυτό θελήσαμε να προωθήσουμε τον ε, οριζόντιο ε, ρόλο που παίζει ο πολιτισμός υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ενταχθεί η πολιτιστική διάσταση στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για το σκοπό αυτό η Προεδρία θα καταθέσει στην Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων ήδη από τη συνεδρίασή της 15 Ιουλίου ένα σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά. Πρόκειται για μια ίδια πρωτοβουλία της Βελγικής Πρωτοβουλίας, την οποία αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία. Θέλουμε με τον τρόπο αυτό να καταλήξουμε σε μια ισόρροπη σχέση ανάμεσα στις τρεις ουσιαστικές διαστάσεις του πολιτισμού, δηλαδή την οικονομική διάσταση, την ε, διάσταση της ηθαγένειας και τη διάσταση της κοινωνικής συνοχής. Θα γίνει ένα συμπόσιο για το θέμα αυτό στις 18 και 19 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες και πάλι. Ο ουσιαστικός ρόλος των δημόσιων βιβλιοθηκών που μπορούν να παίξουν δημόσιες βιβλιοθήκες θα υπογραμμιστεί επίσης στη διάρκεια της Προεδρίας μας και μια, ένα συνέδριο με θέμα η ψηφιακή Ευρώπη και οι δημόσιες βιβλιοθήκες θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό στις Βρυξέλλες στις 20 και στις 21 Σεπτεμβρίου. Τρίτη προτεραιότητα, στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων που έχουν καθαριστεί στον Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πολιτισμού, η Βελγική Προεδρία θα φροντίσει να συμβάλλει στην αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας 2008-2010 για τον πολιτισμό και στην έγκριση ενός νέου σχεδίου εργασίας για την περίοδο μετά το 2010. Διαβάσαμε με ενδιαφέρον τις εκθέσεις κάθε μιας από των 26 χωρών μελών που, που αξιολόγησαν την δουλειά που έχει ήδη γίνει και διαπιστώνουμε ότι όλοι είναι υπέρ της συνέχισης της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού, στο, της μεθόδου ανοιχτού συντονισμού στον τομέα του πολιτισμού, έστω και αν η λειτουργία της μεθόδου αυτής πρέπει να βελτιωθεί ώστε να οδηγεί σε πιο ουσιαστικά αποτελέσματα. Το νέο σχέδιο εργασίας πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να περιέχει πιο επιχειριασιακούς στόχους για σαφώς καθορισμένους συγκεκριμένους τομείς. Πρέπει επίσης να βρεθεί μια καλύτερη σχέση ανάμεσα στις πλατφόρμες, στα, στις, πλαίσια που φέρνουν πιο κοντά την ε, κοινωνία των πολιτών και τις ομάδες εργασίας των εμπειρογνωμόνων. Επίσης η Βελγική Προεδρία θα ορίσει τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν στο πλαίσιο της προώθησης Τη στρατηγική του 2020. Τέλο, η Προεδρία θα συνεχίσει τι συζητήσει που ξεκίνησαν στη διάρκεια τη Ισπανική Προεδρία με σκοπό την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και από, το, την από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της πρότασης απόφασης επιτροπής που έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα σήμα τη Ευρωπαϊκή Κληρονομιά. Με ιδιαίτερη χαρά η Προεδρία θα συνεργαστεί με την κυρία Παλιαντέλη που είναι η συγγήτρια για το θέμα αυτό ώστε να μπορέσουμε σύντομα να καταλήξουμε σε μία συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Η καινοτομία αυτή έχει σκοπό και είναι σημαντικό να μην το ξεχνάμε στι δύσκολε αυτέ περιόδου να φέρει πιο κοντά του πολίτε τη Ευρώπη. Ένα συνέδριο θα οργανωθεί στι 9 Δεκεμβρίου στην Προύζου με σκοπό να συζητηθούν τα μέσα που πρέπει να ε, ληφθούν για να προωθήσουμε αυτή την ευρωπαϊκή στρατηγική της κληρονομιάς. Τώρα, η Προεδρία θα ξεκινήσει μία συζήτηση για τους μηχανισμούς υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Μιλάμε για την πρόκληση της πολιτιστικής πολυμέρειας που κρύβεται πίσω από αυτή την προτεραιότητα. Ο Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος είναι μια από τις καλύτερες εκφράσεις αυτής της πολυμέρειας που μπορούμε να την εγγυηθούμε μόνο εφόσον υπάρξει σημαντική δημόσια υποστήριξη και προώθηση των ευρωπαϊκών έργων. Για το λόγο αυτό οργανώσαμε ήδη από την αρχή της Προεδρίας μας, στις 5 και 6 Ιουλίου στη ΜΟΣ σημαντικό συμπόσιο με σκοπό ακριβώς να σκεφτούμε τα μέσα που θα μας επιτρέψουν να προωθήσουμε την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών ε, ταινιών ώστε να εξασφαλίσουμε την άνθηση της ε, ε, πολιτιστικής περιμέρειας στην Ευρώπη. Το συμπόσιο αυτό έχει ως τίτλο από την ε, οδηγία για, τις, για τα οπτικοακουστικά μέσα στην επικοινωνία κινηματογράφος προς μία σφαιρική και συνεπή προσέγγιση στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο χαρακτηρίστηκε από τεράστια επιτυχία. Συμμετείχαν σε αυτό επαγγελματίες, εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων και εμπειρογνώμων του τομέα, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψει σε εξή θέματα. Πρέπει να υπάρξει δημόσια υποστήριξη σε όλα τα στάδια της αλυσίδα παραγωγή και κυκλοφορία μιας ταινία από τη στιγμή που ετοιμάζεται μέχρι την εκμετάλλευσή τη. Η συνύπαρξη των συστημάτων πολιτιστικής και οικονομικής υποστήριξης μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ισχυρής ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας και ανταγωνιστική συνάμα συμβάλλοντας έτσι στην πολιτιστική πολυμέρεια. Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών και θα θέλαμε να υπάρξει μια άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών ε, των αρμόδιων για, τη, αρμοδίων τη ραδιοτηλεόραση που θα λάβει η χώρα στις Βρυξέλλες την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου ώστε στη διάρκεια αυτής να υπάρξει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα. Ο δεύτερος άξονας εργασίας στον τομέα του, της ραδιοτηλεόρασης εντάσσεται στο πλαίσιο των προκλήσεων που δημιουργεί για όλους μας η ψηφιακή εποχή. Η Προεδρία θα υπογραμμίσει την ανάγκη διαφύλαξης και προστασίας του οπτικοακουστική της οπτικοακουστικής και κινηματογραφικής κληρονομιάς που θα αποτελέσουν αντικείμενο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Η Προεδρία πρέπει επίση να επισύσει την προσοχή του Συμβουλίου στα μέσα που θα χρειαστεί να εφαρμοστούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποστήριξη των αιθουσών κινηματογράφου που θέλουν να εξοπλιστούν με υλικά, υλικό, ε, ψηφιακό υλικό προβολή. Ένα συνέδριο για τι προκλήσει τη ψηφιοποίηση τη οπτικοακουστική κληρονομιά θα γίνει στη Γάνδη στι 13 και 14 Οκτωβρίου. Τέλο, η ανταλλαγή απόψε μεταξύ Υπουργών Λοιπόν στη διάρκεια του επίσημου συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου θα είναι ε, αφιερωμένη σε μια, στη συζήτηση, σε μια συζήτηση για τις πολιτιστικές και οπτικοακουστικές όψεις της, του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Προγράμματος. Σκεφτήκαμε ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό σε επίπεδο Συμβουλίου να προωθήσουμε αυτό το θέμα και τη σχετική συζήτηση, ώστε να μην παραμένει περιορισμένη μόνο στο σχήμα τηλεπικοινωνιών του Συμβουλίου. Οι προοπτικές ανάπτυξης των ψηφιακών βιβλιοθηκών την ψηφιακή εποχή και της Europeana θα εξεταστούν επίσης από την Προεδρία καθώς επίσης και γενικότερες προκλήσεις που θέτει η, διαθέτηση τήρηση σε μακροχρόνιο ορίζοντα του πολιτιστικού, ψηφιακού και οπτικοακουστικού ε, υλικού στην Ευρώπη. Τέλος, η Προεδρία θα οργανώσει 18 Νοεμβρίου μια συνάντηση μεταξύ Συμβουλίου και της Επιτροπής Σοφών με σκοπό που, ε, ε, που, στην οποία έχει ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει συστάσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης, την προσβασιμότητα online και την διαφύλαξη των πολιτιστικών έργων. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μα. Ολοκληρώντα, θέλω να υπογραμμίσω κάποια στοιχεία που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Πρώτον, ε, επιθυμία τη Βελγική Προεδρία είναι να προωθήσει το ψηφιακό πρόγραμμα Επίσης θα προωθήσουμε τον πολιτισμό και τα, τα οπτικοακουστικά μέσα ώστε να μην λειτουργούν πλέον σε στεγανά. Θα πρέπει να δημιουργηθούν γέφυρες και στοιχεία επικοινωνίας με άλλου τομεί ώστε να αξιοποιηθούν πλήρω οι δυνατότητε. Η πρόεδρο τη Επιτροπή σα, η κυρία Ντόρι Πακ, το υπογράμμισε άλλωστε αυτό στην εντυπωσιακή παρέμβαση που έκανε και που ε, προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό στους, σε εκείνους που την άκουσαν στο φόρουμ για τις πολιτιστικές βιομηχανίες που οργανώθηκε από την Ισπανική Προεδρία το Μάρτιο. Το να πούμε ότι πρέπει να εντάξουμε τον πολιτισμό στη στρατηγική 2020 δεν αρκεί πρέπει να πείσουμε τους συναδέλφους των άλλων τομέων και των άλλων κλάδων ότι ο πολιτισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των άλλων δραστηριοτήτων. Η Βελγική Προεδρία σκοπεύει λοιπόν να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη δημιουργικότητα, τον πολιτισμό και την καινοτομία όπως είπα προηγουμένως οι ε, ε, υπεύθυνοι για τα θέματα της ανταγωνιστικότητα του Συμβουλίου πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στο τρίτο θέμα. Σε ό,τι αφορά ε, το, το, το, θέμα της νεολαίας, τον τομέα της νεολαίας, θα επίσης σκοπεύουμε να υπάρξει μια πολύ στενή συνεργασία με το Συμβούλιο έχω κατά νου τα σημεία δημιουργικότητα και πολιτισμός του ψηφίσματος με θέμα η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωσης με σκοπό την επένδυση υπέρ, και ε, ε, των νέων και την κινητοποίησή τους που εγκρίνεται τον περασμένο ε, Μάιο στι 18 Μαου συγκεκριμένα και ο συνάδελφος υπεύθυνο για τα θέματα της νεότητας, ο Πασκάλ Σμέτ, θα παρουσιάσει σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το θέμα της πρόσβασης των νέων στον πολιτισμό. Και οπωσδήποτε θα συνεργαστούμε πολύ στενά μεταξύ μας. Δεν ξεχνάω τέλος την πολιτιστική διάσταση των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια διάσταση για την οποία η στρογγυλή τράπεζα που οργανώσε η πρόεδρό σα, η κυρία Ντόρις Πάξης 23 Ιουνίου, απέδειξε πόσο σημαντική και πόσο πόσο ενδιαφέρουσα είναι. Αυτή η εξωτερική διάσταση θα πρέπει να κατέχει κέρια θέση στο νέο σχέδιο εργασία που ελπίζουμε ότι θα έχει εγκριθεί μέχρι τι 18 Νοεμβρίου από το Συμβούλιο. Σημαντική ημερομηνία, πριν όμω από αυτή την ημερομηνία θα λάβει χώρα η Σύνοδο Κορυφή στη Νέα Υόρκη για τη χιλιετία. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιήσουμε για να εντάξουμε επιτέλου την πολιτιστική διάσταση στου στόχου, στου αναπτυξιακού στόχου τη χιλιετία. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, αυτές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι πεπισμένη ότι μαζί θα εξασφαλίσουμε την επιτυχία, την ουσιαστική επιτυχία της Βελγικής Προεδρίας. Σας ανέφερα τις διάφορες ημερομηνίες για τις οποίες έχουμε προβλέψει μια σειρά από εκδηλώσεις στη διάρκεια της Προεδρίας μας. Βγαίνοντας από την αίθουσα θα βρείτε το πρόγραμμα, το έχετε ήδη έχει μοιραστεί. Σας προσκαλώ σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις λοιπόν και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και περιμένω με ανυπομονησία τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις ερωτήσεις που θα μου υποβάλλετε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Είμαστε στο πλευρό σας αν μας χρειαστείτε. Αλλά πρέπει και εσείς να είστε στο δικό μας πλευρό. Ε? Και αυτό χρειάζεται. Λοιπόν, Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε και στις ε, διασκέψεις, αλλά ξέρετε είναι δύσκολο. Είμαι επιπισμένη όμως ότι αν οι συνάδελφοί μου, αν εγώ δεν μπορώ να είμαι εκεί, θα μπορεί οι συνάδελφοι να εκπροσωπεύσουν την Επιτροπή Πολιτισμού. Σμιτ, δεν ξέρω ποιος. Έχετε σημερομηνίας και αν θέλετε άμα στο το πείτε. Είπαμε στην περίπτωση στην οποία δεν μπορεί να είναι παρούσα η Προεδρία. Ωραία. Έχουν ορισμένοι συνάδελφοι ζητήσει το λόγο. Η κυρία Τσενέσκη πρώτα. Τσενική. Σας ευχαριστώ σε ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα ψηφίσουμε μια έκθεση ε, πολύ σημαντική υπέρ της οποίας θα υπερψηφίσω κι εγώ. Ε, είναι σημαντικό αυτό το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν ξέρω εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα. Με λύπη μου βλέπω ότι οι συναδέλφοι, από άλλες ε, ομάδες ε, δεν καταλαβαίνουν ακριβώ τι θα πει πνευματική ιδιοκτησία. Γιατί από αυτό εξαρτώνται χιλιάδες θέσεις απασχόλησης, μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ. Κύριε Τσανέκη, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα τη Υπουργού εδώ. Ένα άλλο Υπουργό είναι υπεύθυνο για αυτό το θέμα. Κύριε Μπερίκ, είσαι. Δεν θυμάμαι. Α, θα πάει στη Γιούβε, θα πάει στη Γιούβε θα είναι εκεί. Θα το πει και ο Υπουργό. Μπαντίγια. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό γιατί τις τόσο ενδιαφέρουσες και συγκεκριμένες ε, προεδρίες, ε, προτάσεις του προγράμματο τη ε, Βρήκης Προεδρίας. Αναφέρθηκε μάλιστα με τα καλύτερα λόγια στην Ισπανή Υπουργό και θα ήθελα να ευχαριστήσω γι' αυτό. Ελπίζω να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε διάφορα σημαντικά θέματα. Το ένα που με ενδιαφέρει είναι η πράσινη βίβλος για την πολιτική βιομηχανία, για τον πολιτικό κλάδο. Σήμερα ε, το πρωί ακριβώς άκουσα να το θέμα αυτό και ούτε η ίδια ούτε ε, ο εισηγητής αναφέρθηκε καθόλου στο πολιτιστικό τμήμα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Βιομηχανίας για να καταλάβουν ποιο είναι το οικονομικό δυναμικό της του πολιτισμού. Τελειώνοντας, αναφερθήκατε στην πολιτική διάσταση στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον προβλέπεται η κυρία Άστον στο πρόγραμμα εργασίας τη να συμπεριλάβει και αυτό το τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Και αν ναι, πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε μαζί της για τις εξωτερικές σχέσεις. Εγώ έχω διαβάσει το πρόγραμμα της κυρία Σέστον, δεν είχα την εντύπωση ότι ο πολιτισμό θα ήταν ένα θέμα που θα την απασχολήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλοι. Πρόεδρος, Καβαντά. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ένα σχόλιο και μετά δύο ερωτήσει. Το σχόλιο, κύριε Λάναν, είναι να σας πούμε ότι πολλοί βουλευτές και εγώ μεταξύ άλλων δεν φοβούνται και πάρα πολύ την εσωτερική πολιτική κρίση του Βελγίου. Κάθε κράτος έχει την κρίση του. Ο Αναμάρτος λοιπόν πρώτος τον Λίθο Βαλέτο. Εμείς ε, βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ ευρωπαϊκό πνεύμα σε όλες τις διαδοχικές κυβερνήσεις του Βελγίου. Αυτό δεν είναι θα σας καθυσυχάσω. Να μην ανησυχείτε δηλαδή με την εισαγωγή σας εδώ. Οι ερωτήσεις, ερωτήσεις μου είναι αρκετά απλές. Η πρώτη αφορά τον κινηματογραφικό κλάδο στον οποίο αναφερθήκατε. Εγώ είμαι μεταξύ εκείνων που πιστεύουν λόγω μακράς πείρας ότι ένα ευρωπαϊκό ταμείο ευρωπαϊκό λέω, όχι εθνικά ταμεία χρειάζεται απαραίτητα για δύο λόγους γιατί το ευρωπαϊκό πολιτικό κλίμα δεν είναι και καταπληκτικό, αλλά ο πολιτισμό συνεχίζει να δώσει περιεχόμενο. Και δεύτερον, γιατί η ανάπτυξη των ε, ψηφιακών μέσων συμβάλλει πάρα πολύ σημαντικά. Και αυτό είναι το αντικείμενο της δεύτερης ε, ερώτηση για ένα υποσχόλιο μου, κυρία Πρόεδρε. Μου φαίνεται ουσιαστικότατο υπό την Προεδρία σας μια που η πολιτιστική παράδοση στη χώρα αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, κινηματογράφος, ε, ε, κόμιξ, ε, ζωγραφική, αρχιτεκτονική κλπ. Δεν θα σας τα αναφέρω όλο, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν καλό να έχουμε μια ειδική γραμμή για τη δημιουργία περιεχομένου που θα δώσει μια βάση στην ψηφιακή βιομηχανία. Ο πολλαπλασιασμός των διαφόρων διόδων θα βοηθήσει νομίζω. Παλιότερα έγιναν επενδύσεις στον τομέα των, της καλωδιακής τηλεόρασης. Δεν υπήρχε όμως τίποτα για να περάσει από τα καλώδια αυτά και καταστράφηκαν οι επενδυτές. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, ένα ταμείο ή με κοινοτικά φορολογικά κίνητρα ή με άμεση υποστήριξη θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ψηφιακό μέλλον. Γιατί εκτό από τι καθαρές ψηφιακέ υπηρεσίε δεν έχουμε πάρα πολλά θεάματα στον ψηφιακό τομέα και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουν μια ε, δυνατότητα να επιζήσει και να έχει ένα σημαντικό περιεχόμενο. Πρώτος, ευχαριστώ κύριε Καβάντα. Η κυρία Παλιατέλη έχει το λόγο. Ε, θα είμαι πολύ σύντομη. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα ότι ο πολιτισμός τελικά, ακόμη και όταν δεν χρηματοδοτείται τόσο θα έπρεπε, ε, αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο για την Επιτροπή, για το Κοινοβούλιο, αλλά και για τις κυλιόμενες προεδρίες και δηλώνω εδώ πόσο, πόσο μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον, καταθέτω εδώ, πόσο μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον και της Ισπανικής Προεδρίας και της βελγικής αρχόμενης αυτή τη στιγμή προεδρίας σε ό,τι αφορά το σήμα ευρωπαϊκής ε, πολιτικής κληρονομιάς. Ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ε, δώσουμε σε αυτό το σήμα κάτι που ο Βέλγος Πρωθυπουργό ξεκαθάρισε την προχτές στην Ολομέλεια ότι πρέπει να βγούμε πιο επιθετικά τελικά ως Ευρώπη με μεγάλο καμάρι και για την πολιτική μας κληρονομιά. Θεωρώ ότι αυτή η στάση, η επιθετική με την καλή έννοια του όρου είναι ο μόνος τρόπος για να τιμήσουμε πραγματικά μια μεγάλη κληρονομιά στην οποία οφείλεται ίσως ε, ε, αυτό που σήμερα ονομάζουμε δυτικό ε, κόσμο. Να ομολογήσω ότι η Βελγική Προεδρία και ο κύριος Ερικ Πόπε μετέχουν πολύ δυναμικά στην, στις συζητήσεις για το σήμα της πολιτικής κληρονομιάς και να δηλώσω ότι θα ήμουν ευτυχής να τελειώσουμε ε, στην διάρκεια της Προεδρίας της Βελγικής ε, αυτή την συναπόφαση για ένα θεσμό που νομίζω ότι θα συμβάλλει πραγματικά στην ευρωπαϊκή συνοχή και θα δείξει ένα πρόσωπο της Ευρώπης πιο δυναμικό από αυτό που τα τελευταία χρόνια εντοπισμένο μόνο στα οικονομικά κυρίως ζητήματα ε, βρέθηκαν αντιμέτωποι οι προηγούμενες προεδρίες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για όσα μας είπατε. Νομίζω όλοι χαρήκαμε που ήρθατε εδώ και τονίσατε ότι θέλετε η πολιτιστική διάσκεση να ε, παίξει δημιουργικό ρόλο στην ψηφιακή ατζέντα και ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα σας απασχολήσει ιδιαίτερα. Και εγώ θέλω να αναφερθώ στο ψηφιακό μέρισμα. Από ό,τι κατάλαβα θα υποβάλει κάποια σχετική πρόταση η Κομισιόν και ξέρω ότι ακριβώς στον πολιτιστικό τομέα υπάρχουν ακόμα μεγάλα προβλήματα ε, και από εκείνους που προσφέρουν τις υπηρεσίες και που φοβούνται ότι θα φρεθούν στο περιθώριο και από τα θέατρα που φοβούν ότι θα υπάρχει ε, μια επικάλυψη των ε, συχνοτήτων κλπ. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε κάτι σε αυτό, ιδίω να παρακαλέσω την Βελγική Προεδρία και στο ψηφιακό μέρισμα να λάβει υπόψη του ε, το τμήμα αυτό και μας υποστηρίξετε ότι πρέπει να έχουμε τους σωστούς το σωστό επίκεντρο των εργασιών μας, να μην τα αφήσουμε όλα δηλαδή στην πολιτική μόνο, να το πάρουμε και μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής πολιτικής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε την υποστήριξή σας και νύψη της Προεδρίας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τελευταία, η κυρία Γκάλμπετς. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszter asszony, köszönöm szépen az Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Δύο παρατηρήσεις και μια ερώτηση. Πρώτον, έχω δύο παρατηρήσεις που θέλω να κάνω σχετικά με την παρέμβασή Ο πολιτισμός, λέμε, δεν πρέπει να περιθωριοποιείται αυτή είναι μια δήλωση που την άκουσα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Μιλήσατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν στον πολιτιστικό τομέα που θα μπορούσαν να προωθήσουν και να εγγυηθούν την πολιτιστική πολυμέρεια. Συμφωνώ με όλα αυτά. Σε ποιους τομείς όμως ε, έχετε, δίνετε προτεραιότητα στα πλαίσια της δράσης σας. Ευχαριστώ κύριε Μπίσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση που αφορά την ψηφιοποίηση του κινηματογράφου. Με ιδιαίτερη χαρά άκουσα ότι αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στον κινηματογράφο, αλλά υπάρχουν αντιφατικές απόψεις για τον κινηματογράφο. Με την ψηφιοποίηση ο καθένας θα μπορέσει, μπορεί με μια μικρή κάμερα να φτιάξει μια φωτο, να τραβήξει φωτογραφίες, να γυρίσει μια ταινία, ένα ντοκιμοντέρ. Αλλά η ποιότητα των εικόνων ασφαλώς δεν θα είναι τελείως ικανοποιητική. Τι γίνεται λοιπόν με την ποιότητα της, παραγωγικής, της ε, κινηματογραφικής δημιουργίας και παραγωγής. Υπάρχουν ε, αλλαγές που έχουμε διαπιστώσει. Εγώ τουλάχιστον έχω διαπιστώσει σε, πολλές, ε, σε πολλά τηλεοπτικά κανάλια και σε πολλές ταινίε παρατηρείται μία κάμψη, μία μείωση της ποιότητας. Αυτή είναι μια τάση που την έχω διαπιστώσει εγώ προσωπικά και ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Γιατί όταν μιλάμε για πολιτισμό, οπωσδήποτε πρέπει να επιδιώξουμε, να επιδιώξουμε καλύτερη ποιότητα και να τη διαφυλάξουμε. Δεν θέλω να προωθήσω ολυμπιακούς, αισθητικούς ολυμπιακούς αγώνες στον κινηματογράφο. Αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει κάποια ειδική ποιότητα όσον αφορά αυτό το θέμα της παρουσίασης του πολιτισμού στις κάμερες. Πρώτα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα υποβλήθηκαν να μας ρωτήσει στην κυρία Λάνεν. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Euh, euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής σας για το ενδιαφέρον που επέδειξαν για τα θέματα για τα οποία θα είμαι αρμόδια στη χώρα μου αλλά εδώ ως, ε, και εδώ ως πρόεδρος του Συμβουλίου. Και πρέπει να πω ότι οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούσαν την απαγοήτευση που αισθάνεστε εσείς ως ευρωβουλευτές αυτής της Επιτροπής για τα θέματα του πολιτισμού και της ραδιοτηλεόρασης και εγώ βλέποντας ότι αυτά είναι θέματα τα οποία δεν προβάλλονται επαρκώς ενώ όταν συζητάτε με τους άλλους συναδέλφους σας ή με τους δικούς μου συναδέλφους που έχουν άλλες αρμοδιότητες όλοι συμφωνούν ότι ο πολιτισμός είναι μια σημαντική προτεραιότητα αλλά δυστυχώς χρειάζεται κανείς συχνά να αγωνίζεται για να αποκτήσει μερικά πρόσθετα κονδύλια για τον πολιτισμό και να μπορέσει να εντάξει τα θέματα του πολιτισμού σε αποφάσεις και σε νομοθετικά κείμενα και κανονιστικά κείμενα κάτι, μια κατάσταση στην οποία δυστυχώς έχουμε όλοι συνηθίσει. Το ίδιο ισχύει για τις εργασίες που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπουμε στην στρατηγική 2020 ο πολιτισμός δεν περιέχεται σε αυτή τη στρατηγική. Απλώς γίνεται μια προσπάθεια να τον βάλουμε μέσα από την πίσω πόρτα κατά κάποιο τρόπο εντάσσοντάς τον σε άλλες αρμοδιότητες ώστε να προβληθεί κάπως και ο πολιτισμός. Αυτό αντιμετωπίζουμε όλοι μας ανεξάρτητα από τις αρμοδιότητές μας, αλλά αυτό είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει, δεν μας τρομάζει και νομίζω ότι από κοινού θα φροντίσουμε αυτές οι αρμοδιότητες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό να προβληθούν, να προβληθούν και να αποτελέσουν στοιχείο κάθε ευρωπαϊκής πολιτικής. Βεβαίως τρόπο να προβληθούμε, να τραβήξουμε απάνω μας την προσοχή και το ενδιαφέρον. Μιλήσαμε για την πράσινη βίβλο, για τον ε, πολιτιστικό και τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους. Πρέπει λοιπόν να στρέψουμε τους προβολείς πάνω σε αυτό το θέμα που ε, συμβάλλει στην διαμόρφωση και στην ανάπτυξη μιας κοινότητας, μιας κοινωνίας, ενός κράτους και μια ευρύτερης περιοχής όπως είναι η Ευρώπη. Εάν δεν καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα, δεν θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Πρέπει λοιπόν να επαγρυπνούμε, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς θα προβάλλουμε ε, τη σημασία αυτών των κλάδων. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό το τομέα στην Ευρώπη. Που ο τομέας αυτός ε, αντιπροσωπεύει το 2,5% του ΑΕΠ. Η ανάπτυξη των πολιτιστικών κλάδων είναι μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων κλάδων. Όλα αυτά δε και, μπορούμε να δείξουμε ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο, ένα μέσο οικονομικής ανάπτυξης, ένα μέσο που θα επιτρέψει επίσης τη χειραφέτηση του συνόλου των πολιτών. Ένα άλλο σημείο που, ε, στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Παντήλια για την ε, πολιτιστική διάσταση στις εξωτερικές σχέσεις. Πράγματι, στον τομέα της Ευρωπαϊκής υπηρεσ... Ε, διπλωματικής Υπηρεσίας προβλέπεται ότι θα γίνει μια ανάπλαση, αναμόρφωση της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής με την ε, κατάρτιση, κατάρτιση των μελών αυτής της διπλωματικής υπηρεσίας ώστε να προωθούν, να προωθούν τον κλάδο του πολιτισμού, να συνεργάζονται με άλλες χώρες ε, για πάνω σε τομείς που μας ενώνουν. Ο πολιτισμός υπήρξε, ε- η, Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε μαζί με τα κράτη-μέλη τον, ε, την σύμβαση την πολιτιστική σύμβαση της UNESCO. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να βρούμε σημαντικές προσωπικότητες οι οποίες στα πλαίσια των εξωτερικών υποθέσεων θα προβάλλουν τον πολιτισμό σαν ένα μέσο ε, συνεργασίας, αλληλεγγύης, συμφιλίωσης, δεν θα έχουμε φέρει σε πέρα στο έργο μας από πλευράς της κυρίας Άστον, τις επόμενες μέρες θα έχουμε μία ε, επαφή ανάμεσα στις υπηρεσίες μας, ώστε να μας εξηγήσει πώς σκοπεύει να προωθήσει αυτή τη νέα πολιτική που θα αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ παρακολουθώ τις εξελίξεις από πολύ κοντά. Το βλέπουμε σε όλες τις συμφωνίες που υπογράφουμε με άλλα κράτη. Το σκέλος του πολιτισμού είναι πάντα ένα σημαντικό στοιχείο που συμβάλλει ουσιαστικά στις ανταλλαγές μεταξύ εταίρων. Και για να έρθω στις άλλες ερωτήσεις, ο κύριος Καβαντά αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις κινηματογραφικές παραγωγές. Αυτή είναι μια ιδέα την οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική και ενδιαφέρουσα. Η Ευρώπη πράγματι πρέπει να διαδραματίσει σχετικό ρόλο πέρα από τα προγράμματα τα οποία γνωρίζουμε τα προγράμματα των μέσων ενημέρωσης διότι η Ευρώπη μπορεί να συμβάλλει στην πολυμέρεια στην πολιτιστική πολυμέρεια ε, του κινηματογράφου στις διάφορες χώρες. Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος είναι ένας κινηματογράφος που με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με ακτινοβολία παγκόσμια και Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να προωθήσουμε τις κινηματογραφικές παραγωγές. πρέπει να εξασφαλίσουμε υποστήριξη τόσο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να ξεχνάμε ότι στη σκηνηματογραφική παραγωγή η μεγαλύτερη υποστήριξη που παρέχεται από τα κράτη-μέλη συνήθως περιορίζεται στη δημιουργία μιας ταινία. Και ξεχνάμε, έχουμε την τάση να ξεχνάμε ή να είμαστε διστακτικοί, επιφυλακτικοί ίσως λόγω του αισθήματο ότι πρέπει να υπάρξει απόλυτη ελευθερία ανταγωνισμού για τους άλλους τομείς που έχουν άμεση σχέση με τον κινηματογράφο. Όταν ολοκληρωθεί μια ταινία, πολύ ωραία, είμαστε ικανοποιημένοι, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την παραγωγή της, αλλά πριν από την παραγωγή μιας ταινία συμβαίνουν πράγματα, όπως συμβαίνουν πράγματα και μετά την ολοκλήρωση της ταινία. Πρέπει να γίνει διανομή, ε, προβολή, προώθηση της ταινία, να τη γνωρίσουν όλοι οι πολίτες για να την αγαπήσουν όλοι οι πολίτες της Ευρώπης και υπάρχουν μια σειρά από αρμοδιότητες οι οποίες παρεμβαίνουν και χωρίς τις οποίες δεν θα ήταν εύκολη η ζωή των παραγωγών κινηματογραφικών ταινιών. Σκέφτομαι υπάρχουν περιφερειακές ενισχύσεις, φορολογικά κίνητρα για την κινηματογραφική παραγωγή που παρέχονται σε ορισμένες χώρες όπως τη δική μου. Δίνουμε ίσως μια οικονομική διάσταση στο πολιτιστικό προϊόν με αυτόν τον τρόπο, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το απαραίτητο εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε πραγματικά μια ταινία, μια κινηματογραφική και ταινία η οποία θα διαδοθεί και θα τη γνωρίσουν, θα την αγαπήσουν όλοι οι πολίτες της Ευρώπης. Πέρα λοιπόν από την κινηματογραφική παραγωγή χρειάζεται να αναπτύξουμε δραστηριότητα σε όλους αυτούς τους τομείς που ανέφερα. Στη Μόνς, όπως είπα, ε, στην παρέμβασή μου οργανώσαμε ένα συμπόσιο που είχε ακριβώς σαν σκοπό να αναλογιστούμε τις διάφορες μορφές υποστήριξης που μπορούν να δοθούν στην κινηματογραφική παραγωγή χωρίς να περιοριζόμαστε απλά στην παραγωγή μιας ταινίας διότι χρειάζονται αυτές, ε, χρειάζεται μια υποστήριξη και στους άλλους τους τομείς που ανέφερα. πρέπει να επηρεάσουμε τη διαδικασία της ψηφιοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είπατε. Συμφωνώ με τον κύριο Καβαντά και εγώ όταν μας προειδοποιεί λέγοντάς μας ότι δεν πρέπει να εστιαζόμαστε αποκλειστικά στο στην στο μέσο αλλά να δούμε τι θα περάσει, θα διαδοθεί μέσα από αυτό το μέσο. Εσείς ως μέλη αυτής της Επιτροπής είστε ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα, όπως και οι υπουργοί υπεύθυνοι για τη ραδιοτηλεόραση και για τον κινηματογράφο ε, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι ε, για τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την απελευθέρωση και των ε, ΜΜΕ και των νέων τεχνολογιών. Και σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, οπωσδήποτε φορολογικά κίνητρα όπως αυτά που ισχύουν για τον κινηματογράφο θα μπορούσαν να είναι μια λύση Ίσως είναι κάπως πρόωρο αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει μια τέτοια πρωτοβουλία, αλλά οπωσδήποτε θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες ε, διερευνητικές εργασίες ώστε κατόπιν να αναλάβει τη συνέχεια η Ουγγρική Προεδρία που θα διαδεχθεί τη δικιά μας. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα γνωρίζω. Κύριε Παλεντέλη, γιατί έχω ακούσει πολλά για σας και για το ενδιαφέρον, που επιδεικνύεται ε, στα πλαίσια της Επιτροπής για το θέμα με το οποίο ασχολείσαι που είναι το σήμα της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και ελπίζω είναι, συμφωνώ μαζί σου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια διότι μιλάμε για ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρώπη ένα θέμα που θα προβάλλει και θα υπογραμμίζει τη σημασία του να ανήκει κανείς στην Ευρώπη σαν πολίτης σε άμεση σχέση με, με ό,τι όλα τα στοιχεία όλα τα στοιχεία που ακριβώς διαμορφώνουν και δημιουργούν αυτή την Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι πάντοτε μπορεί κανείς να βρει μια λύση, αρκεί να υπάρχει θέληση γι' αυτό. Εγώ ως ε, Βελγίδα ε, είμαι, έχω συνηθίσει στην αναζήτηση συμβιβαστικών λύσεων όπως πολύ καλά το γνωρίζει η κυρία Πακ, ακόμα και παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στο Βέλγιο, ε, πάντοτε καταφέρνουμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση και θα με ενδιέφερε πολύ να ακούσω τις απόψεις σας για κάποια τεχνικά ζητήματα όπως είναι η συμμετοχή των τρίτων χωρών, όπως είναι η μεταβατική διαδικασία και το θέμα ότι ανησυχούμε μήπως υπάρξει ένας πολλαπλασιασμός των τόπων, των τοποθεσιών. Αν έχετε κάποιες ιδέες που θα μπορούσατε να τις μοιραστείτε με την Προεδρία θα είναι ευπρόσδεκτες διότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε να οριστικοποιήσουμε και να ολοκληρώσουμε στη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας. Κυρία Κάμερβερτ, μου υποβάλατε μια ερώτηση για τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή για το θέμα των συχνοτήτων. Ένα θέμα που, που ξέρετε συζητείτε σήμερα και ενδεχομένως να εξελιχθεί σε βάρος των ραδιοσυχνοτήτων υπέρ των ε, τηλεοπτικών συχνοτήτων. Επανέρχομαι λοιπόν και πάλι στο θέμα της ανάγκης προώθησης, με ε, ε, ισομερούς προώθησης των διαφόρων μέσων. Γι' αυτό πρέπει να παραμείνουμε σε στενή επαφή με το Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών συγκεκριμένα, ακριβώ για να αποφύγουμε να μην γίνει μια κατανομή σε βάρο των ραδιοσυχνοτήτων, διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε όλα τα μέσα, όλα τα εργαλεία τη ελευθερία, τη έκφρασης και τη δημοκρατία στις χώρε μα. διότι πολύ συχνά οι, οι τηλεπικοινωνιακές οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών είναι πολύ λέμαριες και προσπαθούν να πάρουν τη μερίδα του λέοντος και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ε, ε, ε, εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια ισομερή κατανομή χωρίς να επιβαρύνεται κανένας. Η κυρία Γκαλπέλτ έκανε μάλλον παρατηρήσεις. Είπατε ότι με χαρά ακούσατε ότι ο πολιτισμός δεν θα βρεθεί στο περιθώριο. Πράγματι μπορώ να σας πω ότι εγώ δεν εγκαταλείπω εύκολα τον αγώνα. Είμαι πολύ αποφασισμένη ε, να κάνω ορισμένα πράγματα, αλλά σέβομαι τις ανταλλαγές με άλλους, τις συζητήσεις ε, τη... και εκεί που, και όταν ε, θα παίρνω το λόγο για να εκφραστώ σας διαβεβαιώ ότι η ραδιοτηλεόραση, ο κινηματογράφος και ο πολιτισμός θα είναι ανάμεσα στα θέματα τα οποία θα υπογραμμίζω και θα προβάλλω. Αυτή είναι η πρώτη επαφή που έχω σήμερα με ευρωβουλευτές για να συζητήσουμε ακριβώς αυτά τα θέματα παρόλο που έχω λάβει μέρος σε άλλες συναντήσεις με την Επιτροπή και τις πολιτικές ομάδες και ποτέ δεν αναφέρθηκαν η ραδιοτηλεόραση, ο κινηματογράφος και τα θέματα του πολιτισμού αυτό με στενοχώρησε πέρα από τις ε, χρηματοπιστωτικές ε, ρυθμίσεις, ε, τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης. Ίσως να φαίνεται ότι ο πολιτισμός είναι λιγότερο σημαντικός, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προβάλλει στην προσωπική και στην κοινωνική ανάπτυξη ο πολιτισμός, αλλά και στην αντιμετώπιση της κρίσης. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να βρίσκεται στο προσκήνιο του ενδιαφέροντός μας. εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι κάποιος που προέρχομαι από πολύ ταπεινή οικογένεια. Ο πολιτισμός, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι ένα μέσο ε, στη διάθεση και εύκολο, στη διάθεση κάθε πολίτη ένα μέσο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης 15% υπάρχουν άνθρωποι των ανθρώπων, των κατοίκων της χώρας μου βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, ένα παιδί στα έξι. είναι κάτι το απίστευτο αυτό την εποχή μας σε μια χώρα όπως το Βέλγιο και υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης αντίστοιχα προβλήματα. Είναι πραγματικά φοβερό να συμβαίνει κάτι τέτοιο και θεωρώ ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει σαν μέσο που θα επιτρέψει στους πολίτες να ξαναβρούν την αξιοπρέπειά τους μέσα τρόπο να αναπτυχθούν, να ανθίσουν σαν άτομα ενώ παράλληλα θα είναι υπεύθυνοι πολίτες, πολίτες που θα ενεργούν και θα συμμετέχουν στη ζωή της κοινωνίας με τη βοήθεια του πολιτισμού. Ποια είναι λοιπόν τα θέματα που κατά την άποψή μου είναι τα πιο σημαντικά. Θα σας πω ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα, ένα θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερα, με το οποίο ασχολούμαι για εδώ και πάνω από έξι χρόνια, εφόσον ε, τα τελευταία έξι χρόνια υπήρξα υπουργό πολιτισμού. Ο κύριος Μπισκή μου υπέβαλε μια κάπως πιο προκλητική ερώτηση, αλλά είναι όμως και μια ουσιαστική ερώτηση για την ποιότητα του πολιτισμού είπε ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα της ψηφιοποίησης και των νέων τεχνολογιών μέσα που πρέπει να φτεθούν ε, στην υπηρεσία του πολιτισμού. Κύριε Μπίσκι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και προσεκτικοί όταν μιλάμε για ποιότητα. Εάν η ποιότητα που εννοείτε εσείς είναι να έχουμε μια πάρα πολύ ωραία αισθητική εικόνα, θεωρώ ότι είναι κάπως επικίνδυνο να χαρακτηρίσουμε έτσι την πολιτιστική παραγωγή, την πολιτιστική δημιουργία. Οπωσδήποτε ε, δίνεται υποστήριξη για τη δημιουργία πραγμάτων που είναι ωραία από αισθητική άποψη. Παράλληλα όμως πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να κάνει πράγματα που να μην είναι απόλυτα ποιοτικά αλλά θα του επιτρέψουν να εκφραστεί καλύτερα. Σε ορισμένα κράτη ε, δίνεται υποστήριξη στον τομέα του κινηματογράφου. Έχω και εγώ εφαρμόσει ένα τέτοιο σύστημα. Έχετε την Επιτροπή Επιλογής των Ταινιών που υποστηρίζει την κινηματογραφική παραγωγή με μεγάλη όπως η αδερφή Νταρντέν. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει ένα ταμείο που υποστηρίζει παράλληλα παραγωγές χαμηλού κόστους που επιτρέπουν σε ταινίε ίσως λιγότερο ενδιαφέρουσες ή λιγότερο ωραίες να παραχθούν διότι αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέσο έκφρασης. Γι' αυτό ε, είναι σημαντικό να έχουμε έργα υψηλής ποιότητας αλλά και έργα τα οποία επιτρέπουν ε, στους πολίτες να βρουν εκεί κάτι που τους, είναι, ε, που τους προσελκύει, κάτι που τους, ε, που τους συγκινεί, κάτι που τους ενδιαφέρει, έστω και αν δεν μιλάμε για μια παραγωγή τεράστιας ποιότητας, της ποιότητας. Κυρία Πακ, ελπίζω ότι απάντησα σε όλους τους παρεμβαίνοντες και τους ευχαριστώ για την προσοχή τους. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, είσαστε πολύ αισιόδοξοι. Είναι μεταδοτικό αυτό και χαίρομαι που έχουμε ζήσει εδώ μια Υπουργό που ξέρει πού είναι τα προβλήματα, ταυτόχρονα όμως δεν εγκαταλείπει την ελπίδα να μπορέσει να ξεπεράσει κάποιο από αυτά. Είναι όπως είπαμε, μεταδοτικό και χαιρόμαστε που σας ακούσαμε σήμερα. Κυρία Πελαδέλη, νομίζω θα πρέπει το γλυγορότερα να ξεκινήσετε να έχετε μια επαφή με την Υπουργό για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό σήμα τη ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Μεταξύ άλλων. Αυτό όμω είναι σημαντικό επίση. Das, was Frau Kammer-Ebert gesagt hat, sehr ernst zu nehmen. Es geht nämlich nicht nur ums Radio. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε θεματικά το θέμα τη ραδιοφωνία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, τα θέατρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μικρόφωνα. Και έχουν ε, την κατάσταση μικρά θέατρα, όπως το δικό μου το θέατρο στο Ζάμπροκεν, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσουν να έχουν μικρόφωνα που να είναι συμβατά με αυτές τις συχνότητες. Δηλαδή, εάν μικρύνουμε ακόμα το φάσμα των συχνοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα θέατρα, θα μειώσουμε τον πολιτισμό μας. Και δεν θα μπορούμε να έχουμε και μεγάλα κονσέρτα στο εσωτερικό των πόλεων. Θα πρέπει όλοι να πηγαίνουν κάπου στην Ήπεθρο για να μην υπάρχουν παρεμποδίσεις από ραδιοφωνικές συχνότητες. Αυτός ο κινδύνος είναι πολύ μεγάλος και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο εάν ε, σμικρύνει ακόμα περισσότερο η ψηφιακή, το ψηφιακό μέρισμα όπως λέμε. Και σας παρακαλώ να το έχετε υπόψη, γιατί αυτό πρόκειται για πολιτισμό για τον καθέναν. Και για κοντσέρτα για αυτούς που τραγουδάνε σανσόν και λοιπά, και για το θέατρο, για την όπερα και όλους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξετάσετε όλα τα θέματα. Δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα. Ε, ε, ε, αναλυτικά θα ήθελα το θέμα Μπίσκι Λάνα να προωθηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς ε, και τους ε, ε, συνεργάτες σας. Ελπίζω να παραμείνετε υπουργό και μετά την δημιουργία της κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ και στο επανειδήν. So, jetzt warten wir auf den nächsten Minister, Pascal Smet.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 Ευχαριστώ. Ο, ήρθε ο Υπουργό. Όλοι οι συνεργάτε ελπίζω να βρήκαν θέση να καθίσουν. Χαίρομαι να σα μπορέσω να σα παρουσιάσω τον Υπουργό για νεότητα ισότητα των ευκαιριών και υποθέσεων τη πόλη των Βρυξελών. Τον κύριο Υπουργό Σμέτ. Είχαμε και μία συνάδελφο που τη λέγανε Σμέτ. Τώρα τη λένε Μάρτεν βέβαια. Αυτό ήταν εκτό ε, το σχόλιο εκτό μικροφόνου. Ε, λοιπόν, χαίρομαι που σα καλωσορίζουμε εδώ. Έχουμε το θέμα της ε, παιδεία. Ένα θέμα που δεν μπορούμε να λύσουμε σε ένα εξάμεινο, αλλά που είναι ένα μόνιμο θέμα, πρέπει να είναι μια μόνιμη μέρημνα. Ελπίζω όμω αυτό το εξάμεινο να μπορέσουμε να έχουμε κάποια ενάβησματα από πλευρά σας Πρόκειται για θέματα κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτισης για νέους, περισσότερο από σημαίνει, τη δυνατότητα απασχόληση, ή απασχολησιμότητα, αν μπορούμε να πούμε έτσι, για τα άτομα αυτά. Ένας από τους στόχους του 2020 είναι να μειώσουμε τον αριθμό εκείνων που εγκαταλείπουν το σχολείο στο 10%, έχουμε υψηλότερη δηλαδή με συμμετοχή εκείνων που έχουν αποβιδίσει από πανεπιστήμια και άλλα παρόμοια ιδρύματα στην Ευρώπη της τάξης του 40% μετά πρόκειται για θέματα νεότητας ε, μείωση της ανεργίας πρόθεση εκείνων των νέων που έχουν κάποια προβλήματα μετανάστες κλπ και όπως ξέρετε έχουμε μια λεγόμενη αγορά εδώ στο σώμα το Νοέμβριο όπου εξετάζεται το θέμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και της επιπτώσεις της στην Ένδια. Πολλά μπορούμε να πούμε, λοιπόν για το θέμα της νότας και μια που εμείς είμαστε όλοι νέοι κινητικοί, όποια ηλικία και αν έχουμε, σας παρακαλώ να μας πείτε κάτι επ' αυτόν. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κύριε Πρόεδρε, και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Θεμάτων, αν εξετάσετε ε, τα θέματα του, ε, του Συμβουλίου Πολιτισμού, θα δείτε ότι έχουμε δύο πολύ σημαντικά σημεία. Αξιολόγηση της διαδικασίας Κοπενχάγης για την ευρωπαϊκή συνεργασία θέματα, σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης ε, που ξεκίνησε πριν από 9 χρόνια στην Μπρίζ ε, που έγινε συνάντηση των Γενικών Διευθυντών που είναι υπεύθυνοι για την επαγγελματική κατάρτιση και στη συνέχεια ένα χρόνο αργότερα το Δεκέμβριο του 2002 υπήρξε για πρώτη φορά η συνεργασία ανάμεσα στους ε, Υπουργούς Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα πάλι εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στη συνέχεια συνέχισε η εργασία αυτή αναπτύχθηκαν νέα ευρωπαϊκά εργαλεία και μέσα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, για τη βελτίωση τη κινητικότητα και τη διαφάνεια. Είχαμε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς ε, Credits. Ε, αυτές ήταν οι πιο σημαντικές ε, μονάδων δηλαδή για τα πανεπιστήμια. Αυτές ήταν οι σημαντικές εξελίξεις. Βεβαίως αυτή τη στιγμή έχουμε την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και η οποία βεβαίω αναπτύσσεται σε κοινωνική κρίση και ελπίζω να μην οδηγήσει και σε κρίση πολιτισμού. Πάντω αυτή τη στιγμή εκατομμύρια άνθρωποι, 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, έχουν πολύ λίγα προσόντα ή καθόλου προσόντα και δεξιότητες. Μέχρι το 2020 θέλουμε να δημιουργηθούν 16 εκατομμύρια θέσει απασχόληση για άκρο ειδικευμένου ανθρώπου, ανθρώπου με υψηλά προσόντα. Αλλά θα μειωθούν κατά 12 εκατομμύρια από ό,τι φαίνεται οι θέσει ανθρώπων, ε, οι ανειδίκευτων ανθρώπων. Ταυτόχρονα γυράζει και ο πληθυσμό, πράγμα που σημαίνει ότι ε, απαιτείται και είναι όλο και πιο σημαντική η συνεχιζόμενη κατάρτιση. Εν ώψη λοιπόν στρατηγική του 2020, και του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση, είναι αλήθεια ότι η επαγγελματική κατάρτιση θα διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο. Έγινε μια συνάντηση το 2004 στο Μάστριχτ και στη συνέχεια το 2006 μια συνάντηση στο Ελσίνκι το και στον Πορντό 2008 και μετά από όλες αυτές τις υπουργικές συναντήσεις θα έχουμε και άλλη μια στην Πρίζα. Ε, από την Πρίζα άλλωστε ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και θα οργανώσουμε στην Πρίζ μια συνεδρία follow-up όπου θα εξετάσουμε το μέλλον. Ε, Στι 6 Δεκεμβρίου του 2010 θα διοργανώσουμε συνδιάσκεψη για την ποιότητα και τη διαφάνεια ω μέσο σύνδεση ε, τη επαγγελματική κατάρτιση και τη εκπαίδευση, ε, σύνδεση των σχολείων και των ε, αντάρτων παστημιακών ε, ιδρυμάτων για ε, να ανοίξουμε δρόμου για την μακροχρόνια ε, τη διαβίου μάθηση. Ε, Μεγάλο ο τίτλο θα μου πείτε τη συνδιάσκεψη. Πάντω σε αυτή τη συνδιάσκεψη θα εξετάσουμε διάφορα ζητήματα, θα εξετάσουμε τη, συνδια της τη ποιότητα, ε, τη αλληλοπερατότητα των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων, τη βελτίωση τη επικοινωνία στου τομεί τη επαγγελματική κατάρτιση κτλ. Πάντω αυτό που σκοπεύουμε να κάνουμε είναι να υπάρξει μία δήλωση, μία διακήρυξη στο τέλο τη διάσκεψη στην Πρίζ ε, όπου θα αξιολογούμε τη συνολική διαδικασία της Κοπεχάγης. Αλλά κυρίως θα εξετάζουμε το μέλλον ε, και θα εκδώσουμε ε, συστάσεις για τις μελλοντικέ προτεραιότητες. Το δεύτερο σημαντικό θέμα στο οποίο θα θέλω να αναφερθώ αφορά την νεολαία σε κίνηση, Youth on the Move. Έχουμε την άτυπη συνεδρίαση, είχαμε την άτυπη συνεδρίαση στη Μαδρίτη, που ήταν η πρώτη φορά όπου υπήρξε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Υπουργών και οι Υπουργοί συζήτησαν ε, το μέλλον και τι ε, θα γίνει στο μέλλον όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό, τι θα συμπεριληφθεί και τι δεν θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα. Και στόχος μας είναι να εργαστούμε με βάση την ανακοίνωση αυτή. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, πολλά να καλύψει όσον αφορά τους ανταγωνιστές μας. Κοιτάξτε, ε, στην ηλικία μου 30-34, λιγότερο από ένα στου τρει Ευρωπαίου ε, έχει πανεπιστημιακό δίπλωμα, ενώ 40% είναι στη ΣΥΠΑ και 50% στην Ιαπωνία. Δηλαδή το 50% των ανθρώπων ε, στην ίδια ηλικιακή ομάδα κατέχουν δίπλωμα πανεπιστημίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενώ της 2020 εμεί θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι ε, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα γίνει πιο ελκυστική, αλλά ταυτόχρονα όχι ει βάρο τη ποιότητα. Εδώ πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στι ευκαιρίε για όλου και στην αριστεία και αυτή η ισορροπία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Λοιπόν, σε αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Όλα αυτά έχουν σχέση με την κινητικότητα, με την απασχόληση, με την αναγνώριση ε, τη ε, επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση. Όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό που θα κάνουμε επί Προεδρία μα είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ, ε, να διοργανώσουμε διερευνητικέ συζητήσει, να προχωρήσουμε όσο μπορούμε, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια προκαταρκτική συζήτηση, μια πρώτη συζήτηση ε, για να δούμε αυτέ τι υποδείξει, τι συστάσει και να δούμε πόσο πολύ μπορούμε μπορούμε να προχωρήσουμε στο προβληματισμό μα. Και βεβαίω αυτό θα εξαρθεί και από τι συνεισφορέ των κρατών μελών και το ε, βαθμό τη συνένεση η οποία θα επιτευχθεί. Όσον αφορά το Youth on the Move, θα διοργανώσουμε μια ευρεία συνδιάσκεψη τον Οκτώβριο. Και βεβαίω θέλουμε να σα καλέσουμε όλου σε αυτή τη διαδικασία. Μιλώ για τι αρχέ τη Οκτωβρίου που θα γίνει η συνδιάσκεψη αυτή. Και για πρώτη φορά σε σχέση με την αηφόρο ανάπτυξη, εμείς θέλουμε το Συμβούλιο να εγκρίνει κάποιε συστάσει. Ξέρετε ότι η αηφόρο ανάπτυξη είναι μια πολύ σημαντική στρατηγική. Και εδώ δεν μιλώ μόνο για την ομοθεσία αλλά για την οτροπία, για την οτροπία των ανθρώπων που πρέπει να αλλάξει. Δεν μιλάω ε, βεβαίω ε, για πλήση εγκεφάλου, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι νέοι Ευρωπαίοι να καταλάβουν, να κατανοήσουν τι μπορεί ε, να τους δώσει η γνώση και οι δεξιότητες και πώς όλα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην βιώσιμη και αηφόρο ανάπτυξη. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ε, θέμα ύψης της σημασίας στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 και είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια του συνολικού ζητήματο τη επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση και τη συνεργασία. Συχνά η αηφόρο ε, ανάπτυξη δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται επαρκώ. Στι 19 λοιπόν Νοεμβρίου ε, θέλουμε να υπάρξουν αυτέ οι συστάσει του Συμβουλίου για τα ζητήματα αυτά τη αηφόρο ανάπτυξη. Γνωρίζετε επίση ότι ένα από τα βασικά προβλήματα στην Ευρώπη είναι το γεγονό ότι πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες, ε, θέματα ε, ε, αλφαβητισμού, γνώσεων βασικών μαθηματικών. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και αποτελούν πρόβλημα για τα παιδιά μας. Επί Γαλλικής Προεδρίας και επί Σουηδικής Προεδρίας υπήρξε σημαντική προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να υπάρξουν κάποιες κατευθυντήρες γραμμές. Υπήρξε κάποια συνεργασία και εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την εργασία. Έγινε ήδη μια συνεδρίαση στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα ακριβώς για τα ζητήματα αυτά. Και όσον αφορά ε, τα παιδιά τα οποία εγκαταλείπουν το σχολείο, εδώ ε, στόχος είναι ένα νούμερο μικρότερο από 10% και θέλουμε ανταλλαγή ευέλικτων πρακτικών. Σε πολλά κράτη-μέλη οι εξελίξει είναι ιδιαίτερα αρνητικέ. Αλλά κοιτάξτε, αν οι άνθρωποι, ε, αν οι πολίτε δεν μπορούν να διαβάσουν καλά, ε, δεν έχουν τι απαραίτητε δεξιότητε, γλωσσικέ δεξιότητε, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν ε, παραπέρα στη ζωή του. Δεν μπορούν να αποκτήσουν υψηλότερη εκπαίδευση και τελικά να ενταχθούν στην αγορά εργασία. Αυτέ είναι ιδιαίτερα αρνητικέ εξελίξει. Και θέλουμε εδώ να κερδίσουμε και να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφο. Να συνεχίσουμε λοιπόν την εργασία τη Γαλλική Προεδρία προ την κατεύθυνση αυτή. Και όπως σας είπα, ήδη έγινε μια συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Και θα υπάρχουν συμπεράσματα του Συμβουλίου και για τα ζητήματα αυτά. Στη συνέχεια, ένα άλλο ζήτημα το οποίο ε, μας ανησυχεί ιδιαίτερα και στις Βρυξέλλες είναι το γεγονό ότι πολλά παιδιά ε, που είχαν ήδη καθυστέρηση όσον αφορά τη μόρφωσή τους και ε, ε, και τα παιδιά τα οποία εγκαταλείπουν το σχολείο πολύ νωρί ή είναι αναλφάβητα, ε, είναι παιδιά μεταναστών. Καταλαβαίνετε ότι τα, προβλήματα, τα παιδιά αυτά κουβαλούν τα προβλήματα αυτά και, στην, και σε ολόκληρη τη ζωή του. Άρα πρέπει να τα βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τα προβλήματα αυτά. Και αυτό είναι και προ όφελο τη κοινωνία συνολικά. Διότι διαφορετικά, αν μου επιτρέπετε να το πω, αν παραμελήσουμε αυτά τα τμήματα του πληθυσμού, η κοινωνία μα θα είναι φτωχότερη. Πρέπει λοιπόν κατά προτεραιότητα να ασχοληθούμε με αυτέ τι πτυχέ τη μετανάστευση. Ε, μετανάστευση δηλαδή σε σχέση με την εκπαίδευση. Ε, και πρέπει να πετύχουμε του στόχου μα στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό έχει να κάνει και με τα σχολεία και με τι περιφέρειες και με, με τι πόλει, όπου υπάρχουν πολλά παιδιά ε, από οικογένειε μεταναστών. Και βεβαίω μιλήσαμε για, το, για, την, για το έτος καταπολέμησης φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού θα διοργανώσουμε μία συνδιάσκεψη το Σεπτέμβριο για την ε, ένταξη στην κοινωνία και θέλουμε να συνεχίσουμε την εργασία μα προ την κατεύθυνση αυτή. Θέλουμε να εξυγχρονίσουμε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και να δούμε πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν επίση πολλά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με του φοιτητέ και τι ανταλλαγέ ανάμεσα ε, στη Γερμανία και στην Αυστρία, ε, στην Γαλλία ε, και στι γαλλόφωνε περιοχέ του Βελγίου. Εκεί όπου υπάρχει έλλειψη αναγνώριση και πρέπει και ισοδυναμία και δυστυχία. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται. όσον αφορά λοιπόν την εκπαίδευση, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αξιολογήσουμε τη διαδικασία της Κοπεχάγης και ίσω αυτό είναι και η βασική μα προτεραιότητα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το μέλλον τη Ευρώπη. Ε, η νεολαία σε κίνηση, πολύ σημαντικό, Η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση επίση. Τώρα δεν μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για τον προπολογισμό του Youth on the Move, αλλά ε, τους προσεχείς μήνες, επί Βελική Προεδρία θα εξετάσουμε με ακρίβεια το πού ε, θα τεθούν οι προτεραιότητές μα και το πώ θα ε, σημειώσουμε πρόοδο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και βέβαια υπάρχει και η φόρο ανάπτυξη, στην οποία αναφέρθηκα. Τέλο, όσον αφορά το μέλλον, το μέλλον της νεολαίας. Κοιτάξτε, αν δεν ασχοληθούμε με το μέλλον τη νεολαία, δεν θα υπάρξει μέλλον για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θα εστιάσουμε την προσοχή μα στην εργασία για του νέου. Το τον Σαββατοκύριακο είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ένα ενδιαφέρον συνέδριο για, ε, για να εξετάσουμε ιστορικά το ζήτημα τη εργασία των νέων και στη συνέχεια είχαμε 350, νεολαίου και εκπροσώπου από τα κράτη-μέλη, από τη Συμβούλια τη Ευρώπη, εμπειρογνώμονε. Όλοι αυτοί συζήτησαν την εργασία ε, για του νέου στην Ευρώπη. Υπήρξε μια διακήρυξη, την οποία νομίζω ότι την πήρατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό, διότι ε, εδώ δεν μιλάμε μόνο για την επίσημη εργασία, αλλά και για τα ανεπίσημα πλαίσια, τα οποία εξίσου είναι σημαντικά, τα άτυπα πλαίσια, η εθελοντική εργασία, ε, ο θελοντισμό, όλα αυτά τα οποία εμπλουτίζουν ε, την ε, ύπαρξή τους και στόχος είναι να υπάρξουν κάποια συμπεράσματα επί Βελικής Προεδρίας, συμπεράσματα ε, για το θέμα αυτό της εργασίας για τους νέους Και πάλι το ξαναλέω, δεν μιλώ μόνο για την τυπική εργασία, αλλά και για τα άτυπα πλαίσια εργασία, τα οποία εξίσου είναι σημαντικά για τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, όταν μιλάμε για τα παιδιά και για τα δικαιώματα των παιδιών, το βασικό τους δικαίωμα είναι το δικαίωμα στο να ε, είναι και να παραμένουν παιδιά. Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο ε, για τη μάθηση ε, και για τα επίσημα σχολικά πλαίσια, αλλά και για το παιχνίδι. Το πώς κανείς μπορεί να μαθαίνει μέσα από το παιχνίδι. Και αυτό είναι σημαντικό. Για να μην παρουσιάζουμε τα πάντα με σοβαρότητα όταν απευθυνόμαστε τα παιδιά. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και θα το, λάβουμε υπόψη και στην περάσμα του Συμβουλίου. Ε, το τρίο των Προεδριών ξεκίνησε ένα δομημένο διάλογο και τις συζητήσεις με το ε, ε, European Youth Forum και με την κοινωνία των πολιτών. Όλα αυτά θα τα συνεχίσουμε και ε, θα προετοιμάσουμε την εργασία μας προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και όλα αυτά θα κορυφωθούν στις συστάσεις, όπως σας είπα. Ένα άλλο θέμα που έχει προτεραιότητα στην ατζέντα μας είναι τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων ανθρώπων. Ήδη έχει γίνει σημαντικό μέρος εργασίας αυτής Έχουμε τη Σύμβαση των Ηνωμένων για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Συνθήκη τη Λισαβόνα. Όλα αυτά τώρα πρέπει να συγκεντρωθούν. Και εμεί ε, έχουμε την εντύπωση ότι πολλά γίνονται στο συγκεκριμένο τομέα. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη σύγκληση, περισσότερο συντονισμό. Ε, να αντιλήσουμε ε, προσθέμενη αξία από τη συνέργεια και να λάβουμε υπόψη όλε τι προσπάθειε. Και θα, θα διοργανώσουμε μια συνδιάσκεψη και για το θέμα αυτό. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θα διοργανώσουμε. Ε, μία εκδήλωση εδώ στις Βρυξέλλες, στην πρωτεύουσα της Ευρώπης, για την νεολαία στην Ευρώπη στις 27 Νοεμβρίου και είστε όλοι προσκεκλημένοι. Πρόκειται για μία εκδήλωση όπου θα συγκεντρωθούν νέοι εδώ στην Ευρώπη για να δουν το πώς τα παιδιά και οι νέοι μπορεί να συμμετάσχουν ε, στα τεκτενόμενα στην πόλη, στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, ένα στου δύο ε, ε, ανθρώπου που μένει στι Βρυξέλλε δεν γεννήθηκε ο ίδιο ή οι γονεί του στι Βρυξέλλε. Και σε 20 χρόνια ε, οι 7 στου 10 ε, κατοίκου των Βρυξελών ε, δεν θα είναι ε, βελγική καταγωγή. Κοιτάξτε, και από τη δική μου προφορά καταλαβαίνετε ότι και εγώ δεν είμαι βρυξελιώτη, ε, γέννημα θρέμα. Πάντω αυτή η τάση ε, θα ενταθεί στο μέλλον. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε πολλέ προκλήσει να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να τι ε, δούμε αυτέ και να τι δούμε επί βελγική προεδρία. Και ταυτόχρονα θέλουμε να προσπαθήσουμε να ε, πετύχουμε ε, ανταλλαγή απόψεων ε, σε επίπεδο νεολαία. Κοιτάξτε, εγώ ω αρμόδιο υπουργό τη Βρυξέλλε χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ε, είμαι υπεύθυνο και για την νεολαία και για την παιδεία. Είναι πολύ σημαντική η διασύνδεση των δύο θεμάτων. Αυτό σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε για το μέλλον. Ε, εφτά συνάδελφοι συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνοι και για τα δύο θέματα, και εκπαίδευση και νεολαία. Καταλαβαίνετε ο, λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να κάτσουμε ε, όλοι μαζί και να πετύχουμε ένα είδος ε, ε, ε, συντονισμού όλων αυτών των τομέων πολιτικής. Γιατί μερικές φορές υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στην εκπαίδευση, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την εκπαίδευση και την νεολαία. παιδεία μερικές φορές σημαίνει τι δεν μπορούν να κάνουν οι νέοι. Ενώ οι νέοι χρησιμοποιούν λέξεις όπως εθελοντισμό, για παράδειγμα, που σημαίνει τι μπορούν να κάνουν. Πρέπει λοιπόν να γεφυρώσουμε όλε αυτέ τι πτυχέ. Αυτό θα το κάνουμε λοιπόν επί Βελική Προεδρίας. και είμαι σίγουρο ότι θα έχω να σα πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα για πρόοδο συγκεκριμένη στο τομέα. Αυτέ λοιπόν οι προτεραιότητέ μα, αυτέ οι προτεραιότητε τη Βελική και σας λέω ότι έχουμε μεγάλο ενθουσιασμό, ξεκινήσαμε μεγάλο ενθουσιασμό και ελπίζω να συνεχίσουμε όλοι με τον ίδιο ρυθμό και με τον ίδιο ενθουσιασμό. Σε τελευταία ανάλυση αυτό το πρόγραμμα είναι κάτι που μας αφορά όλους. Όπω και, όπως και η προηγούμενη συνάδελφος είπε, είμαστε πολύ καλοί εμεί στο Βέλγιο ε, στον τομέα των συμβασμών. Έχουμε παράδοση. Βλέπουμε την ευρύτερη εικόνα και αυτό κάνουμε και στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Πολλά είπατε. Πολλά σκοπεύετε να κάνετε. Ξέρετε ότι είσαι δεσμευμένη σε μια τριπλή προεδρία, σε μια τρόικα. Πολλά από αυτά δηλαδή που έχετε κατά νου, που θέλετε να ξεκινήσετε, θα μπορούσαν να συνεχίσουν στην επόμενη προεδρία. Αυτό είναι το πολύ καλό στην πρόθεση, ότι δεν περιοριζόμαστε μόνο σε ένα εξάμεινο, μπορεί κανένα να προβλέψει καλύτερα στο μέλλον. Ωραία. Μία σειρά συναδέλφων έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ, έστε όλοι σύντομοι και υποβάλλετε ερωτήσει. Ο κύριο Φέρα, από τη Σλοβενία. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ε, κύριε Υπουργέ, πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση των προτεραιοτήτων σας. Ήταν πολύ καλές και ε, μερικές φορές ε, δημιουργείται η εντύπωση ότι ε, τελικά ε, έχουμε καλύψει τα πάντα και ότι καμία προεδρία δεν μπορεί να είναι πρωτότυπη. Ότι δηλαδή τα πάντα έχουν ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν μπορεί κανεί να κάνει τίποτα το καινούριο. Όμω, ε, νομίζω ότι με, σωστή, με το σωστό ενθουσιασμό, ρυθμό και ενέργεια μπορεί, μπορούν οι διάφορε προεδρίε να δώσουν έμφαση σε διάφορα θέματα που αφορούν την νεολαία και την εκπαίδευση. Και τώρα που αρχίζω να γνωρίζω τους Βέλγους υπουργού, νομίζω ότι όλοι είστε ιδιαίτερα ικανοί και όλοι ε, διακατέχεστε από ιδιαίτερη ε, δημιουργικότητα ε, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τα θέματα που μας απασχολούν. Εσείς αναφέρατε τη διαδικασία της Κοπενχάγης για την επαγγελματική κατάρτιση. Και ίσως θα έπρεπε να τονίσουμε όχι μόνο τη δευτερογενή επαγγελματική κατάρτιση, αλλά την επαγγελματική κατάρτιση γενικά. Ε, είχαμε ε, διάφορα ε, έχουμε διάφορα γενικά γυμνάσια και λύκεια, και λύκεια που, που προετοιμάζουν και αυτά το, τους νέους για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Και όμως εκεί είναι το πρόβλημα και όχι τόσο σε επίπεδο επαγγελματική κατάρτισης γιατί αυτά τα σχολεία ε, παρέχουν γενικές δεξιότητες στους νέους και είναι ακόμα πιο δύσκολο για αυτούς στη συνέχεια να ενταχθούν στην αγορά εργασία. Λοιπόν, φαίνεται ότι η μοναδική δυνατότητα είναι να συνεχίσουν ε, τις σπουδέ τους σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και θα ήθελα να σα πω το εξή: Το 2008 ήταν ε, το έτος του διαπολιτισμικού διαλόγου. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους ασχοληθήκαμε με το διαπολιτισμικό διάλογο, με τις γλώσσες, ε, επί γερμανικής, ε, ε, σλοβενικής προεδρίας κλπ. Δημιουργήθηκε μια ιδέα, υπήρξε μια ιδέα για κάποιους δείκτες αξιολόγησης της γνώσης της δεύτερης και τρίτης ξένης γλώσσας των νέων. Αυτό είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, γιατί Η πίεση εκ των έξω μπορεί να δώσει νέα όθηση κίνητρα ε, στα εθνικά συστήματα παιδείας και να αποτελέσει το κίνητρο για την διδασκαλία ξένων γλωσσών να το νωρίτερα. Και ίσως αυτό είναι μια ιδέα που θα πρέπει να αναβιωθεί και θα μπορούσε να, γίνει, να γίνουν περισσότερα προς την κατεύθυνση αυτή. Και τελειώνω να σα κάνω μια ερώτηση. τελειώνοντα λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μία σειρά από πρωτοβουλίε. Μία από αυτέ είναι αυτό το θέμα το Youth on the Move, τη νεολαία εκκίνηση, που αναφέρατε κι εσεί. Είναι πολύ ευρία η πρωτοβουλία αυτή και σίγουρα υπάρχουν ορισμένε πτυχέ και ορισμένα προγράμματα που Ίσως θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε άλλα προγράμματα, όπω για παράδειγμα το πρόγραμμα διαβίου, διαβίου μάθησης που έχει και ευρύτερη ε, χρηματική υποστήριξη. Ποια είναι η άποψή σα, λοιπόν όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ε, δεχθούμε αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή να προτείνουμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά τα δύο αυτά προγράμματα. Uh, uh, uh, Herr ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την εισαγωγή αυτή που μας κάνατε, κύριε Υπουργέ, και σας εύχομαι κάθε επιτυχία το επόμενο εξάμεινο. Συμφωνούμε νομίζω πάνω σε πολλά από αυτά που παρουσιάσατε. Αλλά έχω μία ερώτηση στην διαβίου μάθηση. Α, εμείς είμαστε πάρα πολύ διασμεσμένοι με τη διαδικασία της Βολόνια. Έχουμε δηλαδή 20% φοιτητών στο πρόγραμμα Εράσμους μέχρι το 2020. Τα τελευταία χρόνια είχαμε ήδη 10%. Αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά δύο πράγματα θα πρέπει να σκεφτούμε. Αυτοί οι στόχοι δεν θα πρέπει να αποδυναμωθούν. Γιατί οι ορισμένοι λένε ε, ότι 20% για το 2020 ε, θα ήταν πολύ καλό να έχουν ε, οι φοιτητέ ε, εμπειρία από το εξωτερικό. Αυτό αφορά όμως μόνο ένα τμήμα της εκπαίδευσής τους. Δηλαδή, εάν οι μαθητές και οι φοιτητές πάνε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, καλό είναι. Τι γίνεται όμως με την ανώτατη εκπαίδευση να μην υπάρχει αποδυνάμωση και το θέμα του προπολογισμού επίσης για την διαβίου μάθηση το Συμβούλιο πρότεινε να περικοπεί το σχετικό κονδύλο κατά 25 εκατομμύρια ευρώ και ο εισηγητής μας του Κοινοβουλίου είπε ότι αυτό είναι μια πραγματική πρόκληση και συμφωνούμε μαζί του. Γιατί εάν ένα πρόγραμμα υπάρχει πάνω στο οποίο θα πρέπει να, να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε για το μέλλον, ακριβώ η διαβίου μάθηση. Πρώτα σας ευχαριστώ κύριος Παπενικολάου. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και πράγματι είναι ενθουσιώδης η προσέγγιση που μας κάνατε. Ε, πράγματι είναι φιλόδοξος ο προγραμματισμός σας. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε ενημερωθεί ότι στον προσεχή προϋπολογισμό στα θέματα παιδείας και στα θέματα που αφορούν τους νέους θα έχουμε σημαντικές περικοπές. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση της δικής σας Προεδρίας σε αυτό. Το δεύτερο, είναι πολύ σημαντικός ο προγραμματισμός ό,τι αφορά τις συναντήσεις που θα διοργανώσετε, τις διασκέψεις ε, για συγκεκριμένα θέματα. Μήπως είναι ευκαιρία αυτές οι πρωτοβουλίες να συνδυαστούν και με τα προβλήματα που όλοι διαπιστώνουμε, το είπαμε και την προηγούμενη, στην προηγούμενη ε, συνάντηση της Επιτροπής μας με την απελθούσα Ισπανική Προεδρία και τον ομόλογό σας από την Ισπανία. Μήπως πρέπει να δούμε και τα προβλήματα της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού και παράλληλα με τις συναντήσεις αυτές που θα διοργανώσετε να έχουμε και κάποιους υπότιτλους ε, και να επεξεργαστούμε προτάσεις και λύσεις για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Γιατί το έχουμε ξαναπεί και νομίζω φαίνεται αυτό και στο σχεδιασμό που έχει το Συμβούλιο και η Επιτροπή, το είπαμε και εμείς στην έκθεσή μας για τους νέους. Εμείς εδώ λέμε πολλά και σημαντικά, η αφομοίωσή τους όμως στα κράτη-μέλη δεν είναι αυτή που πρέπει. Θα είναι πολύ σημαντική η συνδρομή της Βελικής Προεδρίας, αυτή είναι η δική μου άποψη, αν με αυτές τις πρωτοβουλίες που ήδη έχετε εξαγγείλει μπορέσουμε να δούμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε για τον συντονισμό και την αφομοίωση των πολιτικών που χαράσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς όπως γνωρίζουμε η επικουρικότητα δημιουργεί σημαντικές δυσχέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Παντία. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Υπουργό για τις εξηγήσεις του σχετικά με τις προτεραιότητες σε θέματα εκπαίδευσης και νεολαίας και θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, διαδικασία στην αξιολόγηση διαδικασία τη Κοπενχάγη, στην οποία αναφερθήκατε. Για μένα αυτή είναι μια από τι πιο σημαντικέ προτεραιότητε, ίσω η πρώτη προτεραιότητα μεταξύ όλων αυτών που αναφέρατε. Αλλά έχω κάποιε αμφιβολίες για, σχετικά με αυτό που σκοπεύετε να κάνετε. Τα είδαμε τα προβλήματα, τα κατανοήσαμε τα προβλήματα που οδήγησαν στη διαδικασία της Μπολόνια σε πολλές χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να αντλήσουμε διδάγματα από τα προβλήματα αυτά τα οποία οδήγησαν στη διαδικασία της Μπολόνια. Και στα πλαίσια της διαδικασίας Κοπενχάγης δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε το παρελθόν. Συμφωνώ με τους άλλους ευρωβουλευτές όταν προσπαθώ να εξηγήσω το περιεχόμενο της διαδικασίας της Κοπενχάγης χωρίς να ξέρει κανείς την αυτή διαδικασία στη χώρα μου. Ερωτώ λοιπόν, όταν μας λέτε ότι προβλέπονται συνεδριάσεις που γίνονται κάθε δύο χρόνια μέσα από τις οποίες γίνεται αξιολόγηση διαδικασίας Κοπενχάγης. Ποιοι συμμετέχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις. Όταν μιλάμε για τη διαδικασία της Μπολόνια, ξέρουμε ότι ήταν οι εκπρόσωποι των πανεπιστημίων που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις. Εδώ όμως μια και μιλάμε για κατάρτιση μιλάμε για επιχειρήσεις, για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης. Πρέπει να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει την αξιολόγηση και την προώθηση της δυναμικής της διαδικασίας της Κοπενχάγη και θα έπρεπε οι περιφέρειες να παίζουν πιο σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία για να την προωθήσουν. Ευχαριστώ κυρία Μελίτα Λόβα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, άκουσα με προσοχή αυτά που μας είπατε και πραγματικά ε, με εντυπωσίασε το ότι είσαι τόσο αποφασισμένος και τόσο ενθουσιώδης. Από την άλλη μεριά όμως μου έλειψαν κάποια συγκεκριμένα βήματα που θέλετε να κάνετε. Δεν άκουσα τίποτα για την υποστήριξη της νεολαίας, δεν άκουσα τίποτα για την πολιτική για την νεολαία συγκεκριμένο και για την παιδεία της νεολαίας συγκεκριμένο. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης το θέμα της απασχόλησης της νεολαία είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η ανεργία μεταξύ των νέων είναι 20%. Και αυτό είναι κάτι λοιπόν που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και αυτό που είναι επίσης σημαντικό κατά τη γνώμη μας είναι να υποστηρίξουμε την επαγγελματική κατάρτιση γιατί νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα κενά και να μην αναφερόμαστε πάντα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση αλλά και στην επαγγελματική κατάρτιση. Και αυτό χρειάζεται. Και έχω να σας πω επίσης ότι μου αρέσει πάρα πολύ η πρωτοβουλία αυτή η νεολαία η Youth on the Move. Και πάνω σε αυτό έχω να πω ότι κατά τη γνώμη μου όλοι προσπαθούμε να προωθήσουμε κάποια νέα ταξινόμηση πανεπιστημίων Ίσως αυτό να είναι μια υποραπλούστευση των προγραμμάτων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω ίσως να ε, περιορίσουμε την προσοχή μας στην βελτίωση της ποιότητας των πανεπιστήμιων ούτως ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν άλλα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Θα ήθελα να ξέρω τι θέλετε να κάνετε πάνω σε αυτό. Και πώς, πώς δηλαδή θα βελτιώσετε την ποιότητα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ο συνάδελφος Μπόρις έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για τις δηλώσεις σας. Μας έπαιρνε με μεγάλο ενθουσιασμό, πολλή ενέργεια Θα ήθελα να σε την προσοχή μας ε, στα κύρια στοιχεία της στρατηγικής του 2020. Το μια κατά 10% αύξηση εκείνων που έχουν πανεπιστημιακή κατάρτιση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, η αύξηση εκείνων που έχουν επαγγελματικά ε, επαγγελματικές κανόνες. Το 1 τρίτο των νέων δεν έχουν τέτοια, ε, τέτοια επαγγελματικά προσόντα. Άκουσα προσεκτικά αυτό που είπατε, ότι ξεκινάτε σε μια άκουσα στην οποία θα πρέπει να συνεχίσουν οι επόμενε προεδρία. Συγκεκριμένα όμως τι σκοπεύετε να κάνετε για να μπορέσουν οι δύο αυτοί οι δείχτες να βελτιωθούν. σκοπεύετε να δράσετε ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί μέσα στα πλαίσια των ε, νέων δημοσιονομικών προοπτικών για να βελτιωθεί η επαγγελματική κατάρτιση και οι Υπουργοί παιδεία των κρατών μελών θα μπορέσουν να εμπλακούν εδώ για να βελτιωθούν και να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Πρόεδρο, συνάδελφοι, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε ακόμα τέσσερι που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα κάνω μια διακοπή για να μπορέσει ο υπουργό να απαντήσει στα πιο σημαντικά θέματα. Δέκα λεπτά το πολύ και μετά οι επόμενοι συνάδελφοι. Δεν χρειάζεται να επαναλάβετε όλα όσα είπατε Καμιά φορά δεν πρόσεχαν καν οι συνάδελφοι και έχουμε διπλά, διπλές τις ερωτήσεις. Λοιπόν, το πολύ 10 λεπτά για τι απαντήσεις και μετά θα συνεχίσουμε. Αλλιώ θα είμαστε άδικοι. Παρακαλώ, Υπουργό, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι ακόμα πιο σύντομο. Συμφωνώ για, σχετικά με τη διαδικασία της Κοπενχάγης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η διαδικασία αυτή να μην περιλαμβάνει μόνο τους φοιτητές αλλά και τους μαθητευόμενους. Και αυτοί όλοι να έχουν καλές γνώσεις μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, συμφωνούμε. Ακόμα καλύτερα και δύο ξένων γλωσσών και πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη διαδικασία της Μπολόνια αλλά και τη διαδικασία της Κοπενχάγης. 32 χώρες παραπάνω από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ε, οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλοι κάθονται γύρω από το τραπέζι. Το ξέρετε ίσως και υπάρχει μια παράδοση την παραμονή του Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας γίνεται μια άτυπη συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους και την Προεδρία της ε, Τριμερούς Ομάδας, του Τρίο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε πραγματικά δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο σε αυτή την άτυπη συνάντηση. Είναι ενδιαφέρον το ότι γίνεται αυτή η συνάντηση, αλλά πρέπει να έχει και ουσιαστικό περιεχόμενο. Αυτή λοιπόν η άτυπη συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους, εμείς θα προσπαθήσουμε να εστιαστεί σε μια ουσιαστική συζήτηση για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, την, την εκπόνηση προγραμμάτων μαθητείας και μάθηση ώστε για να μπορούν τα άτομα να περνάνε από τη μία εκπαίδευση και μια κατάρτιση σε μία επόμενη και να προχωρήσουν κατόπιν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ε, αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία σε όλα αυτά. Ε, τώρα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιφέρειες. Ως Βέλγος υπουργό ε, θα πω βεβαίως ναι, ως, υπουργός του, πρόεδρος του Συμβουλίου θα πω αυτό θα το αποφασίσει κάθε κράτος μέλος μεμονωμένα πώς σκοπεύει να προωθήσει δηλαδή αυτή τη διαδικασία. Όταν όμως ζούμε σε μια ομοσπονδιακή χώρα με περιφέρειες οι οποίες έχουν τι ε, δικέ δικές, τις δικές τους αρμοδιότητες είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία ώστε να πετυχαίνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και, πρέπει σε ορισμένες ε, περιπτώσεις να εμπλακούν στην όλη διαδικασία και οι κοινότητες να υπάρχει ένα σύνδεσμος ανάμεσα σε όλα αυτά τα επίπεδα για να κινούμαστε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση, να καταβάλουμε προσπάθειες για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Το πρόγραμμα Youth, η πρωτοβουλία Youth on the Move, η νεολαία ε, σε κίνηση, στην άτυπη συνάντηση, στο άτυπο συμβούλιο έγινε μια, μια εκτεταμένη συζήτηση για το τι ακριβώς καλύπτει αυτή η ονομασία. Είναι μια διαφορετική ονομασία για το πρόγραμμα διαβίου μάθησης. Όταν μιλάμε για το πρόγραμμα διαβίου μάθησης, δεν μιλάμε μόνο για τους νέους, αλλά και για τους ενήλικες. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση αν ενταχθούν στο πρόγραμμα Youth on the Move και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό και οι ενήλικες από πλευράς επικοινωνιακής θα υπάρξουν προβλήματα, οπωσδήποτε δεν είναι το συμπέρασμά μου αυτό, αλλά είναι αυτή η κατεύθυνση που έδωσε αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξει σαφής διαχωρισμός. Όταν μιλάμε για το πρόγραμμα Youth on the Move, μιλάμε μόνο για τους νέους. Δεν λέμε ότι δεν είναι σημαντική η διαβίου μάθηση, οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Θα περιμένουμε βεβαίω την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε ποιε είναι οι θέσει τη. Πάντω, εγώ στην ανακοίνωση αυτή πιστεύω ότι δεν μιλάμε μόνο για κινητικότητα, για ποιότητα τη εκπαίδευση, αλλά ότι υπάρχει και ένα κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στην απασχόληση και στην ανεργία των νέων και δεν ε, ε, ε, υπάγεται στην αρμοδιότητα ενός μόνου επιτρόπου. Γι' αυτό θα δούμε πώς θα βρούμε την καλύτερη δυνατή ισορροπία για να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Ο στόχος του Συμβουλίου είναι να είμαστε σε επαφή και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια σε βάθο συζήτηση για το θέμα αυτό. Οι στόχοι είναι σημαντική στη στρατηγική Ευρώπη 2020 πρέπει να μεταφερθούν κάποιοι ευρωπαϊκοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο. Αυτή θα είναι μια σημαντική προσπάθεια και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για τη χώρα μου δεν μπορούμε να πούμε ότι θα αναπαυθούμε στις δάφνες μας. Χρειάζεται ακόμα να γίνει πολλή δουλειά. Αν δούμε το, τις ομάδες των μεταναστών, δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Χρειάζεται να γίνει ακόμα πολλή δουλειά και αυτό ασφαλώς ισχύει και σε άλλες χώρες. Επίσης πρέπει να δούμε πώς θα αξιολογήσουμε, θα μετρήσουμε τα αποτελέσματα στα πλαίσια της εθνικής εμπειρίας. Ε, αν πάρουμε τους δείκτες, ε, μπορεί να έχουμε πετύχει τους στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε μεμονωμένες χώρες, όπως στην ε, Φλαμανδία παραδείγματο χάρη, στην περίπτωση της Φλάνδρας, στη φλαμανδική περίπτωση, οι στόχοι, οι δείκτες αυτοί δεν έχουν καλυφθεί. Βεβαίως ε, βλέπουμε για να δούμε, για να δούμε ε, ακριβώς τι πρέπει να γίνει, πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στο προπολογισμό. Διότι χωρίς προπολογισμό, χωρίς αρκετά κονδύλια, δεν ωφελεί να γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση. Οι Υπουργοί Παιδείας ομόφωνα ε, στη Μαδρίτη είπαν ότι όλα αυτά πρέπει να μεταφραστούν, να, μεταφραστούν σε κονδύλια. Θα χρειαστεί λοιπόν να γίνει μια σημαντική προσπάθεια και αυτή τη στιγμή δεδομένης της ε, οικονομικής ε, συγκυρίας μιλάμε για 20,5 ε, εκατομμύρια ευρώ για το 2011 για τον προϋπολογισμό της, του προγράμματος της διαβίου μάθησης πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η διοικητική διαχείριση του προγράμματος, ποια θα είναι τα επιμέρους έργα, ποια είναι τα ποσοστά υλοποίησης, τι έγινε, τι πραγματοποιήθηκε και τι δεν πραγματοποιήθηκε ακόμα, τι δεν υλοποιήθηκε ακόμα. Υπάρχει μια πρόταση στο τραπέζι αυτή τη στιγμή όπως ξέρετε, έχετε ενημερωθεί σχετικά. Ομιλώ λοιπόν ε, εξ ονόματος των Υπουργών Παιδείας εμείς λέμε ότι καλύτερο θα ήταν να μην γίνονταν οικονομίες, αλλά ε, δυστυχώς θα χρειαστεί να βρούμε μια ισορροπία, διότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα που χρειάζονται χρηματοδότηση. Αλλά συμφωνούμε μαζί σας ότι πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ε, και αυτό ισχύει για την πολιτική. Όταν λέμε ότι η παιδεία, η εκπαίδευση είναι σημαντική, πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη στα επιμέρους προγράμματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Περιφερειακό Ταμείο θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επαγγελματικής κατάρτισης. Θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό στο μέλλον. Και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, διότι βλέπω να μου κάνετε νόημα ότι πρέπει να σταματήσω, η ποιότητα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το, το θέμα. περιλαμβάνεται στο, στη δικασία της Μπολόνια. Βρίσκεται ίσως κάπως εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα από τα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Σε άτυπο επίπεδο θα δούμε πώς ε, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά υπάρχει αυτή η αξιολόγηση, η κατάταξη, χρειαζόμαστε μία κατάταξη ε, των ε, Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, υπάρχουν υπέρ και κατά. Θα προχωρήσουμε λοιπόν, θα μελετήσουμε το θέμα για να δούμε πώς προοδευτικά, με συνεπή και ρεαλιστικό τρόπο θα βρούμε τα κατάλληλα, τα σωστά κριτήρια, διότι πρόκειται για δύσκολη προσπάθεια και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν προβαίνουμε σε συγκρίσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η πρώτος εκτό μικροφώνου όμως. Σας παρακαλώ, επόμενη συνάδελφη, πάρα πολύ σύντομη. Φύσες. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήδη πολλέ από τι ερωτήσει που θα μπορούσα να υποβάλω με καλύφθηκα από του προηγούμενου και, το, και τα απάντησε πολύ σωστά ο Υπουργό. Δύο θέματα θέλω να πω. Το πρώτο αφορά την κινητικότητα των καθηγητών στα πλαίσια τη διαδικασία τη Μπολόνια. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα Ερασμού σε επίπεδο νέων ήταν πολύ πετυχημένο πρόγραμμα, αλλά νομίζω ότι ε, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε όσον αφορά την κινητικότητα των καθηγητών μέσα στην Ευρώπη ε, στα πλαίσια τη διαδικασία Μπολόνια. Και δεν ξέρω αν υπήρξε σημαντική πρόοδο. Επίση, μιλήσατε για τα προβλήματα ε, που μπορεί να υπάρξουν ε, ανάμεσα ε, στο πρόγραμμα της διαβίου μάθησης και, και στην κινητικότητα των νέων, στα δύο προγράμματα. Κοιτάξτε όμως, αυτή τη στιγμή το μέλλον πολλών ανθρώπων σε μεγαλύτερη ηλικία στην Ευρώπη, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν πρόσβαση στη νέα τεχνολογία κτλ. και στους υπόλοιπους. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι η νεολαία βεβαίως είναι σημαντική, αλλά μην ξεχνάμε και τους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους και τη σημασία που έχει το πρόγραμμα αυτό και για αυτούς. Ευχαριστούμε. Κυρία Κώστα έχει το λόγο. Θα σε ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ ε, τον Υπουργό για, αυτό το, ε, για αυτά που μας είπε για το πνεύμα με το οποίο αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό. Είναι στρατηγική σημασία ε, περισσότερη σύνδεση τη πολιτική παιδεία και τη πολιτική υπέρ των νέων. Και αυτό και για ένα ακόμα λόγο που έχει να κάνει με το χαμηλό ε, προφίλ ε, της συνθήκης Λισαβόνα στα ζητήματα αυτά και στην κοινοτική αρμοδιότητα. Ε, οι νέοι στα πλαίσια της συνθήκης Λισαβόνας αναφέρονται ότι είναι ε, ε, πρωταγωνιστές ε, των πολιτικών. Θα πρέπει μάλλον να είναι πρωταγωνιστές και όχι μόνο να είναι δικαιούχοι όλων αυτών των πολιτικών, να δέχονται τις πολιτικές. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, έχουμε το άρθρο 166 της συνθήκης καινοτομία. Εκεί προβλέπεται ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει πέραν της, του σεβασμού της αρχής επικουρικότητας, που βεβαίως την ξέρουμε στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει όμως να βρουν τα κατάλληλα μέσα και μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ε, Σα παραπέμπω και εγώ σε αυτά που είναι συνάδελφοι και ίσω η στρατηγική 2020 στον τομέα αυτό δεν έχει ε, ακόμα ε, προσδιορίσει την απαραίτητη αναθεώρηση των μέσων ε, της διακυβέρνησης και του ελέγχου. Ε, αναφέρονται μόνο στόχοι, χωρίς όμως να σταθούμε για λίγο και να δούμε γιατί μέχρι στιγμής δεν έγινε τίποτα με τους στόχους αυτούς. Διαφορετικά δεν θα κάνουμε τίποτα. Τελευταίο, όσον αφορά το μέτωπο της διαδικασίας Κοπεχάγης. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο ε, αν ε, σε κάποια από τις πρωτοβουλίε σας, και εγώ πιστεύω ότι αυτό κάνετε, θα μπορούσατε να δείτε όχι μόνο πού βρισκόμαστε ε, όσον αφορά το σύστημα των προσόντων κτλ, αλλά να δείτε ποιε είναι οι βέλτιστε πρακτικές, ποιε είναι οι πιο πετυχημένε πρακτικές. Ε, ε, και ε, με αυτόν τον τρόπο να αναφέρονται συγκεκριμένε υποδείξει το 2020. Διαφορετικά αναφέρονται αριθμητικοί στόχοι, χωρί όμω να συνοδεύονται και από μια στρατηγική που μπορεί να μα οδηγήσει στόχου αυτού. Κυρία Σάκη. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, minister. Um, hartelijk dank voor uw ambitieus. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, Υπουργέ, σας ευχαριστώ για τόσο βιλόδοξο πρόγραμμά σας που προβλέπει πραγματικά και ταινίζει προς το μέλλον. Ορισμένα νόμματα δεν αναφέρθηκαν. Όταν μιλάει κανένα για την νεολαία και το μέλλον, θα πρέπει να έχει κατά νου την ψηφιακή ατζέντα, την ανάπτυξη τη σύγχρονη τεχνολογία που έχει σημαντικέ επιπτώσει στου νέου. Σε όλου μα, αλλά στου νέου ιδιαίτερα. Γιατί πραγματικά μεγαλώνουν σε διαφορετικού καιρού. Ε, όσον αφορά τα νέα ΜΜΕ και τη χρήση των νέων μέσων στην ε, παιδεία, τι έχετε κατά νου, έχουμε το διαδίκτυο, υπάρχει όμως και η σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων, ανθρώπων που έρχονται από μετασ... Ε, οικογένειες μεταναστών, άλλους. Ποια είναι τα διάφορα προγράμματα που έχει η Ευρώπη που ξεπερνάνε τα σύνορα όσον αφορά την παιδεία, την νεολαία και τον πολιτισμό. Εγώ θα προετοιμάσω μια σχετική έκθεση το φθινόπωρο και θέλετε μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα από κοινού. Ακριβώς. Πολιτισμό, νέα μέσα και ιστορική ε, πολιτική Η κυρία Χόνιμπολ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ τον Υπουργό. Το να αποκαλείται αυτόν υπουργό του μέλλοντος είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί αυτό που αρχίζει να είναι προβληματικό είναι η παιδεία στις μικρές ηλικίε. Γιατί άμα θέλουμε να έχουμε καλύτερη ένταξη στην κοινωνία, καλύτερες επαγγελματικές ε, ικανότητες, θα πρέπει να αρχίσουμε πραγματικά στην αρχή της ηλικίας των παιδιών, της ε, παιδείας των παιδιών. Και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον η Βελική Προεδρία έχει κάποια σχέδια προς την κατεύθυνση αυτή. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος τελειώσαμε. Πέντε λεπτά έχουμε ακόμα. Το πολύ. Γιατί ο συνάδελφό σα είναι έξω από την πόρτα. Όχι για μένα, για τον συνάδελφό σα που είναι έξω από την πόρτα και περιμένει. Άμα αυτό έχει τον αθλητισμό. Α, ε, δεν πειράζει. άστιο αστείο ήταν. Θα του πω μόνο, μόνο αθλητισμό. Θα του το πω. Κοιτάξτε, είναι ισπανικής, ε, ισπανικής καταγωγής και είναι πολύ ευτυχισμένος αυτές τις μέρες. Δεν τον πειράζει λοιπόν τίποτα. Και εγώ αυτή είμαι, εγώ είμαι ένα υπέρ τη Ισπανίας. Ε. Ε, και τι να σα κάνω εσάς εδώ. Λοιπόν, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Ε, όσον αφορά την κινητικότητα των καθηγητών. Ναι, έχετε δίκιο. Ξέρουμε ότι υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα όταν συζητάμε για την ε, νεολαία εγκινήση. Είπαμε ότι θα εξετάσουμε την Τράπεζα Επενδύσεων και με το Συμβούλιο και την Κομισιόν να δούμε πού μπορούμε να βρούμε νέες πηγές χρηματοδότησης ούτω ώστε και οι φοιτητέ και οι καθηγητές να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αυτές τις ε, ανταλλαγές στο εξωτερικό. Θα το εξετάσουμε λοιπόν γιατί είναι δύσκολο. Συμμετοχή των νέων, ναι, συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτό ακριβώς προωθούμε αυτό τον διαστρωμένο διάλογο που ξεκίνησε με την Ισπανική Προεδρία και μάλιστα ίσως και πριν από αυτήν να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Ε, οι νέοι και η εργασία υπάρχει το φόρουμ της Νορέας, υπάρχουν εθνικές ε, ο, επιτροπές που αξιολογούν κάποιον διαρθρωμένο διάλογο, θα γίνει και στην Ουγγρική Προεδρία αυτή, για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συσχετισμός. Προσωρινή αναθεώρηση στρατηγικής 2020. Ναι, όλοι οι συνάδελφοι και με τον συνάδελφο στην όταν πάει στη Μαδρίση συμφωνήσαμε, ε, συμφωνήσαμε ψηφιακή ατζέντα. Κύριε Χάκερ, συμφωνώ, δεν έχουμε άμεσα ε, σχέδια. Θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των συνεδριάσεων. Δεν έχουμε όμως συγκεντρώσει την προσοχή μας, αλλά ευχαριστώ να το συζητήσουμε το θέμα. Ε, παιδεία, πολιτισμός, μετανάστευση. Το Σεπτέμβριο, νομίζω είχε προανακριθεί αυτό στη Στοκόλμη, ε, έχει αναδειχθεί μια μελέτη για τη στάση των νέων και των παιδιών όσον αφορά την ενεργή συμμετοχή στη δημοκρατία και στα του κράτους. Πολλοί νέοι δεν είχαν ίσως πολύ επιτυχείς εμπειρίες εδώ. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό να εξάσουμε συζητήσεις. Να ευχαριστώ. Θαυμάσια, θαυμάσια λέει η πρόεδρος. Καλό δεν ήταν. Ναι, πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καταπληκτικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Πάρα πολύ ευχάριστα αυτά. Είδαμε έτσι πολύ ωραίους και ευχάριστους υπουργού εδώ. Είμαι πολύ ευτυχής που ε, αφιερώνει τόσο πολύ ενέργεια η Βελική Προεδρία σε αυτά τα θέματα. Τη χρειαζόμαστε, γιατί ακριβώς σε αυτό το τομέα βρίσκεται η ψυχή της Ευρώπης. Αν δεν επενδύσουμε εκεί, χάσαμε. Μας τα είπατε και πολύ καλύτερα από ό,τι σας το λέω εγώ σήμερα. Και γι' αυτό θα ήμουν ε, ευτυχής εάν η Βελική Προεδρία και στις συναντήσεις των υπουργών μπορέσει να δώσεις μια μεγαλύτερη όθηση και να ρωτήσει τον καθένα τι κάνατε εσείς. Πρέπει κανένας να πιέσει αυτούς να εργαστούν. Όταν ο ένας λέει ναι εγώ έκανα αυτό και αυτό και αυτό, ο άλλος δεν έχει να πει τίποτα, ίσως την επόμενη φορά θα έχει τη φιλοδοξία να παρουσιάσει και εκείνος κάτι προς όφελος των παιδιών μας και των παιδιών των παιδιών μας. Πρέπει λοιπόν πολλά να κάνουμε. Έχετε εσεί τα σωστά ενάβμασα. Έχουμε εμπιστοσύνη σε εσά και ελπίζουμε το επόμενο εξάμεινο να μπορέσετε να εκκινήσετε κάποια πράγματα που να μπορούσαν να συνεχιστούν στην επόμενη Προεδρία και ίσω και να ολοκληρωθούν. Αλλά βέβαια νομίζω ότι θα είναι αιώνια εργασία πάνω σε αυτό το θέμα. Είσαστε λοιπόν ένα κρίκο στην αλυσίδα, αλλά νομίζω πολύ απολυσματικό. Καλή τύχη, σα ευχαριστώ που ήρθατε. Λοιπόν, είχα τελείως ξεχάσει το θέμα του παγκοσμίου κυπέλου και να συγχαρώ τους Ισπανούς. Συγχαρητήρια στους Ισπανούς. Αλλά και οι Ολλανδοί έπαιξαν καλά, ε? εντάξει. Και οι Γερμανοί που πήραν την τρίτη θέση. You did not play? What? <laughs> Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. You disagree. You disagree. Διαφωνείτε. Διαφωνείτε. Γιατί διαφωνείτε. Πιστεύετε ότι πραγματικά έπαιξαν δίκαια και σαν gentleman οι Ολλανδοί. Εγώ δεν είπα δίκαια, είπα καλά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, ξεχάστε το. Ω, πάπα, πάπα, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση γιατί δεν θα βγούμε να έρθουμε σε αυτό τον Υπουργό που είναι μόνο, μόνο για τον αθλητισμό, όπως είπε ο συνάδελφός του. Χαίρομαι λοιπόν που είναι εδώ παρόν ο Υπουργό Αθλητισμού. Μια πρώτη φορά έχουμε την δυνατότητα μετά τη Λισαβόνα. Ξεκινήσαμε με την Ισπανία, αλλά μετά τη Λισαβόνα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με κάποιον που μπορεί να ε, ξεκινήσει τα θέματα. Hm, Χαιρόμαστε λοιπόν που ο Υπουργό Ιωσμίτε είναι εδώ και μπορεί να μας πει τι πρόκειται να κάνει τα επόμενα χρόνια. Η Κομισιόν μας είπε ότι στις 10 Νοεμβρίου θα υποβάλει μια πρόταση για ένα διετές ε, πρόγραμμα μέχρι το 2013 για τον αθλητισμό και θα τη δείξουμε εμπιστοσύνη ότι θα είναι καλό το περιεχόμενο, μπορείτε ακόμα να συμβάλλετε σε αυτό και ότι θα έχουμε και περισσότερα χρήματα. Γι' αυτό δεν είναι υπεύθυνη η Κομισιόν. Θα πρέπει να βασιστεί και στη δική σας υποστήριξη όπως και εμείς. Δεν μπορούμε να έχουμε τον αθλητισμό τώρα στη συνθήκη και στις ιδέες αυτές για τα επόμενα δύο χρόνια να μην δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα από εκείνα που δαπανούσαμε όταν δεν είχαμε αρμοδιότητα. Αυτό θα ήταν πραγματικά ανέκδοτο. Λοιπόν, παρακαλώ, μας παρουσιάσετε τις προτάσεις σας. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Eh, ε, Κυρίε και κύριοι μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού, κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Βελικής Προεδρίας για τον αθλητισμό. Και βεβαίως ε, με πολύ μεγάλη μου χαρά να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις σας. Στο παρελθόν είχα διαβάσει ιδιαίτερα τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό και ξέρω πόση μεγάλη σημασία αποδίδεται στον αθλητισμό. Έχετε εκδώσει ψηφίσματα, έχετε κάνει συνεδριάσεις, ε, επιτροπές υψηλού επίπεδου. Έχουν γίνει πολλά για το θέμα του αθλητισμού. Ξέρω λοιπόν τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό. Και αυτός ο ενεργός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήδη ξεκίνησε με την έκθεση ΠΑΚ το 1997 δείχνει το πόσο σημαντική είναι η ε, πολιτική σε θέματα αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω όλα αυτά ε, οδήγησαν στη συνθήκη τη Λισαβόνα, εκεί όπου ε, αναφέρεται, αναφέρονται συγκεκριμένε αρμοδιότητε του Κοινοβουλίου σε θέματα αθλητισμού. Και αυτέ είναι ιδιαίτερα θετικέ εξελίξει. Αυτή η νέα νομική βάση είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς ως Βελική Προεδρία χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε εδώ ε, με την αρχή αυτής της νέας εποχής για την πολιτική αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω ότι επί Βελικής Προεδρίας να συμβάλλουμε ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα αθλητισμού. Φυσικά ε, υπάρχει μια ανακοίνωση για τα ζητήματα αυτά. Και με αυτή τη βάση θα ξεκινήσουμε την εργασία μας. Έχουμε διάφορες προτεραιότητες σε θέματα αθλητισμού. Πρώτα απ' όλα το πλαίσιο ε, για τι ε, πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μελλοντικέ πολιτικέ και για το ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία, συμπεριλαμβάνοντα και το fair play. Αυτά είναι ε, τα δύο βασικά ζητήματα. Όσον αφορά το μέλλον των πολιτικών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ περιμένουμε με ανυπομονησία αυτή την ανακοίνωση και τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμά τη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και η συνθήκη τη Λισαβόνα δημιούργησε σημαντικές προσδοκίες και στον τομέα του αθλητισμού αλλά και στα ίδια τα κράτη-μέλη. Και πρέπει να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα ως προς τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα του αθλητισμού. Τι κατεύθυνση πρέπει ε, να ακολουθήσουμε. Στο Συμβούλιο συζητήσαμε στις 10 Μαΐου το ζήτημα αυτό και βλέπω ότι οι προσδοκίες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Πρόεδρε, ε, αναφερθήκατε σε διάφορες ε, ε, πολιτικές σε θέματα αθλητισμού. Εμεί οι Προεδρίε μα θα ε, συγκεντρώσουμε την προσοχή μα στα ζητήματα αυτά. Έχουμε δομένο διάλογο με τον, τομέα, και με τον κλάδο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και υπάρχει συνένεση γύρω από το ποιο θα συμμετάσχει στο διάλογο αυτό. Ο προκατοχό μου, ε, εκ μέρου Ισπανία, έκανε το πρώτο βήμα όσον αφορά την επίτευξη συνένεση με, ε, με του τομέα στη, ε, προς τη συμμετοχή στο δεμένο διάλογο, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα μία σειρά πρακτικά ζητήματα. Τον τρόπο εργασίας, την ημερήσια διάταξη, πρακτικά ζητήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω. Ο δεμένος διάλογο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα ζητήματα αυτά. Και βεβαίω δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα των συζητήσεων, αλλά θα ήθελα να σα πω ότι η Βελική Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη επίσημης απόφασης εκ μέρους του Συμβουλίου. Με τη μορφή ψηφίσματος ελπίζουμε. έτσι ώστε να ξεκαθαριστούν αυτά τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκα. σε διάταξη, πρακτικές ε, ε, δυσκολίες, ε, λεπτομέρειες εργασίες κτλ. Το δεύτερο τώρα θέμα το οποίο, στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ο ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία. Συμπεριλαμβάνοντα και το εφαγωνίζεστε, το fair play. Και εδώ υπάρχουν διάφοροι υποτομεί. Η, η κοινωνική ένταξη ε, στον, το, στον τομέα του αθλητισμού και από τον αθλητισμό, ή ε, ο αθλητισμό και η κατάρτιση και το πώς ε, αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν για να καταπολεμήσουμε ε, τα, το, το ντοπάρισμα. Επίσης πρέπει να δούμε πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός. Και αυτή τη στιγμή απευθυνόμαστε και στην επόμενη Προεδρία της Ουγγαρίας και την Προεδρία της Πολωνίας για να δούμε πώς μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Για τα τρία τώρα υποθέματα στα οποία αναφέρθηκα. Βεβαίω ήδη ξέρουμε ότι το 2010 είναι το ευρωπαϊκό έτο για την καταπολέμηση τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και αυτέ οι προτεραιότητε σίγουρα θα συνεχίσουν και στην ε, επόμενη Προεδρία. Υπήρξε το Λευκό Βιβλίο για τον Αθλητισμό, που υπογραμμίζει το θετικό ρόλο του αθλητισμού και οι προπαρασκευαστικές δράσεις που ήδη έχει αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2009 αλλά και για το 2010 που εξακολουθούν να θέτουν ως προτεραιότητα τον αθλητισμό. Νομίζω ότι ε, αν εξετάσουμε ε, το εφαγωνίζεστε, τη συναδελφικότητα, τον αθλητισμό, τη δέσμευση, την επικοινωνία, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά και πρέπει να εξετάζονται από κοινού με το θέμα του αθλητισμού. Γιατί εδώ σε τελευταία ανάλυση μπορούμε να δούμε το ρόλο του αθλητισμού ε, στην κοινωνία. Να σας πω ότι στο παρελθόν ήμουν προπονητής ε, ε, ε, ομάδας νέων και είχα δει με πρώτο, πρώτο χέρι το πώς ε, εκεί ε, έρχονται ε, και συνεργάζονται άνθρωποι με χαμηλά προσόντα από ταπεινά κοινωνικά στρώματα και έρχονται σε επαφή και με τους υπόλοιπους και όλοι μαζί εργάζονται και συνεργάζονται μέσα σε ένα θετικό κλίμα. Επιτόπου μπορεί κανείς να δει τη θετική επίδραση του αθλητισμού στην κοινωνία από πρώτο χέρι. Και βεβαίω μπορείτε να δείτε τα θέματα τη κατάρτιση και τη εκπαίδευση. Αλλά εδώ μιλάμε ε, για πτυχέ εκτό σχολείου που είναι εξίσου σημαντικέ. Οι νέοι μπορούν να μαθαίνουν με διάφορου τρόπου. Και νομίζω ότι ο αθλητισμό είναι ε, μια απο τι πολυ θετικε μορφε μαθηση πολύ θετική πτυχή ε, που θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα έχει να κάνει με τη διοργάνωση μια συνδιάσκεψη για την κοινωνική ένταξη. Θέλουμε λοιπόν ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στου εμπειρογνώμονε για να δούμε πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Πάλι με θέμα το θετικό ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία. Εδώ βεβαίω δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τον τροχό, αρκεί να αντλήσουμε από τη θετική εμπειρία που ήδη υπάρχει. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία στα οποία θέλουμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μα επί Βελική Προεδρία. Κάτι άλλο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το εξή. Θέλουμε κάποια συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα θέματα κοινωνική ένταξη σε συνδυασμό του αθλητισμό. Βεβαίω, ε, αυτό, σε αυτό ήδη αναφέρθηκα. Αλλά τώρα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Το, τον αθλητισμό και την κατάρτιση. Και πώ μπορούμε να προωθήσουμε αυτέ τι πτυχέ σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να έχουμε ε, καλή κατάρτιση για τον αθλητισμό αλλά και καλή προπόνηση αν θέλετε ε, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Πλαισίου ε, Απόκτηση Προσόντων στον τομέα του αθλητισμού έχουμε το θέμα ε, της διπλής σταδιοδρομίας και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μπορεί ε, κάποιοι άνθρωποι να ασχολούνται με τον αθλητισμό αλλά και με άλλες μορφές κατάρτισης. Ε, Βεβαίω υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ε, αθλητέ ε, που κερδίζουν πολλά από τη δραστηριότητά του. Αλλά τι γίνεται μετά όταν αποσυρθούν, ε, πώ συνεχίζουν την καριέρα του. Γι' αυτό μιλώ για ε, ε τη, τη δυτή καριέρα. Και βέβαια και το θέμα ε, τη πληρωμή των νέων κατά τη διάρκεια ε, τη κατάρτιση και τη προπόνηση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Και εδώ πρέπει να αλλάξουμε απόψει. Και σίγουρα αυτό θα γίνει επί Βελική Προεδρία, θα ανταλλάξουμε απόψει. Κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και προκύπτει διαρκώ είναι η καταπολέμηση του ντόπινγκ. Η νέα νομική βάση για τον αθλητισμό εστιάζεται ε, στην προστασία ε, της ε, σωματικής και ηθικής ακαιρεότητας των αθλητών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ισχυρότερο ρόλο. Ζητώ συγγνώμη, ε, ε, έχουμε παρεμβολέ από τα κινητά. Ε, διακόπτη πρόεδρο. Συνεχίζω, λέει ο μιλητή. Ε, πανέρχομαι λοιπόν στο θέμα του ντόπινγκ. Στην Ευρώπη έχουμε πολλέ χώρες ή περιφέρειες που έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή του κώδικα της WADA. Και ακριβώς γι' αυτό ε, γι' αυτό εμείς αναθέσαμε ε, μία ε, μελέτη από το Ινστιτούτο Άσερ για να δούμε ποιοι εφαρμόζουν, ποια κράτη-μέλη εφαρμόζουν και πώς εφαρμόζουν τον κώδικα αυτό ε, της WADA. Δηλαδή, μερικές φορές τι γίνεται. Ένα πράγμα είναι η συγκεκριμένη νομοθεσία και ένα άλλο το πώ εφαρμόζεται και υλοποιείται. Θέλουμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά στι λεπτομέρειέ του και είναι πολύ σημαντικά. Να δούμε και τι διαφορέ που υπάρχουν όσον αφορά την ε, πρακτική εφαρμογή του κώδικα αυτού της ΓΟΑΝΤΑ. Θα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα επί Βελικής Προεδρίας. Και όλα αυτά θα αποτελέσουν μια καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις. Και στα πλαίσια της ΓΟΑΝΤΑ. Ε, ε, υπάρχουν άνθρωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ε, ΓΟΑΝΤΑ και μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη είναι ένα μικρό τμήμα και μόνο τη Ε, Εμεί δηλαδή ε, παίζουμε μικρό ρόλο, αν θέλετε. Και μερικές, εκεί και μερικέ φορέ είναι και δύσκολο να ακουστεί η φωνή μα. Όσον αφορά λοιπόν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα, εδώ ε, βλέπουμε τα πράγματα από τελείω διαφορετική σκοπιά από ότι πολλέ ε, άλλε χώρε που συμμετέχουν σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ουάντα. Η προστασία λοιπόν της, του ιδιωτικού απορρίτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο προβλέπεται και συνταγματικά σε ορισμένα κράτη-μέλη, προβλέπεται και από το Σύνταγμα. Και να σας πω ότι το Μάιο πήγα εγώ ε, στη Γουάντα και έκανα κάποια σχόλια προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά ήταν κάπως παράξενη η, η αντίδραση που συνάντησα. Του είπα ότι αυτό είναι αντισταγματικό και μου είπαν «Ε, τότε αλλάξτε το, αναφέρω στο σύνταγμά σα. Ε, μα είναι απάντηση αυτή. Άρα λοιπόν ε, πρέπει ε, να, να ακουστεί η φωνή μα ε, ε, ισχυρότερα. Γιατί η φιλοσοφία μα είναι διαφορετική και θα πρέπει να την προωθήσουμε αυτή τη φιλοσοφία μας Έχουμε την UNESCO, έχουμε το Συμβούλιο τη Ευρώπη, όλους αυτούς τους φορείς που θα πρέπει να εμπλακούν εδώ στη συζήτηση και θα πρέπει να εξετάσουμε το πώ μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων. σω λοιπόν θα μπορούσα να σταματήσω εδώ, αναφέροντα και ορισμένε εκδηλώσει συγκεκριμένε που θα διοργανωθούν επί Βελγική Προεδρία. Ε, πάντα για το τομέα του αθλητισμού. Πρώτα απ' όλα θα το ξέρετε, 18 και 19 Νοεμβρίου έχουμε το Συμβούλιο Παιδεία και Νεολαία. και ο αθλητισμός θα συζητηθεί το απόγευμα τη 18 η Νοεμβρίου. Μετά θα έχουμε την άτυπη συνεδρίαση την άτομη συνεδρίαση με τους συναδέλφους μου, τους ομολόγους μου, στην Αμβέρσα, 21 και 22 Οκτωβρίου. Αλλά ε, προηγουμένω 16 και 17 Σεπτεμβρίου θα συναντηθούν οι διευθυντέ ε, σε, σε, σε, θέματα αθλητισμού και μετά γίνουν δύο συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων που θα διοργανωθούν και σα καλώ και εσά. Ε, η πρώτη θα γίνει, θα ασχοληθεί με θέματα κοινωνική ένταξη και θα συζητήσουμε στους ε, ε, τοπικούς πολιτικούς, σε αυτούς που χαράσουν πολιτικές και θα αντλήσουμε συμπεράσματα και διδάγματα από τις βέλτιστες πρακτικές. Και επίσης έχουμε και την Ευρωπαϊκή ημέρα των προπονητών. Ε, αυτό το διοργανώνουμε στη Φλάνδρα κάθε δύο χρόνια. εκεί όπου γίνεται η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους προπονητές ε, υψηλού επίπεδου. Θα το ξαναδούμε λοιπόν αυτό, αλλά θέλουμε, ε, θα το ξανακάνουμε λοιπόν αυτή τη διάσκεψη, αλλά θέλουμε να είναι ευρωπαϊκή εκδήλωση αυτή τη φορά και να ε, κάνουμε ανταλλαγή απόψεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πολύ καλή η συνεισφορά μας. Αυτό, είναι ορισμένα τα πράγματα που θέλω να πω για πολύ. Ευχαριστώ. Οκτώ, οκτώ συνάδελφοι, εφτά. Α, πόσοι, δύο, τέσσερις, έξι, οκτώ. Οκτώ, εννέα, εννέα. Ο, ο καθένας από ένα λεπτό, εντάξει. Σύνομη και επί της ουσίας. Η κυρία Μποσκότ. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, minister, voor uw uh, inleiding. Oh. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τη δήλωσή σας. Θα ήθελα να πω ξεκινώντας ότι σέβομαι απόλυτα την, προεδρική, την Βελγική Προεδρία. Έχετε πάρα πολλή δουλειά να κάνετε. Θέλετε να αντιμετωπίσετε το θέμα της φαρμακοδιέγερσης και την ρυθμίσεις που έχει προβλέψει η ΟΑΝΤΑ θα ήταν καλύτερο νομίζω να εκπροσωπείται πιο αποτελεσματικά και πιο, με πιο ολοκληρωμένο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση στον, στη Ουάντα. Μιλήσατε για τη μελέτη του Ινστιτούτου σχετικά με την εξολόγηση των διαφόρων μέτρων υπάρχει το θέμα του άρθρου 29 θα ήθελα λίγο περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό κοινωνική ενσωμάτωση για, για, και για τους ποδοσφαιρικές ομάδες και για τους αθλητικούς ε, μήλους νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι προωθούν την κοινωνική ενσωμάτωση και μπορούν να ζητήσουν ε, ε, χρηματοδότηση αλλά πολλές φορές οι υπεύθυνοι που διαχειρίζονται αυτά τα ταμεία δεν έχουν αντιληφθεί ότι είναι σημαντικό να συμπεριλάβουν μεταξύ των αποδεκτών των κονδυλίων τους και τους αθλητικούς ομίλους. Ευχαριστώ. Η Βελγική Προεδρία πράγματι μας παρουσίασε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία. Χωρίς χρήματα τίποτε όμως δεν μπορεί να γίνει. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και ως εισηγητής για τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, εγώ διαπίστωσα ότι τα ποσά που προβλέπονται για τον ε, για να στηρίξουν αυτή την νέα πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ περιορισμένα Νομίζω ότι ομιλώ εξ ονόματο όλων λέγοντα ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ένα πιο σημαντικό προπολογισμό ώστε να ενισχυθούν πραγματικά όλες αυτές οι πρωτοβουλίε τις οποίε υποστηρίζουμε. Δεύτερη ερώτηση. Στην ομάδα συζητήσαμε με τον ε, Επίτροπο για το θέμα αυτό. Μια και μιλάμε για το, την κοινωνική πτυχή Μήπως θα μπορούσαμε να οργανώνουμε ευρωπαϊκά τουρνουά στα σχολεία, τουρνουά ποδοσφαίρου στα σχολεία. Στη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας θα είσαστε έτοιμος να αναλάβετε μια τέτοια πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Κύριος Φίσας, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε για τα συγχαρητήριά σας. Πρέπει να σας πω ότι ε, είδαμε μαζί ε, τον αγώνα κατά της Γερμανίας και εσείς πρόεδρε ήταν οι πρώτοι που ήρθατε και μου δώσατε συγχαρτήρια για την ε, νίκη μας τότε. Ευχαριστούμε Υπουργέ. νομίζω ότι η σύνοψή σας είναι πληρέστατη και καλύψατε πολλά θέματα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να είμαι σύντομο, δεν μπορώ να μιλήσω για πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι. Αλλά θα ήθελα να, να τονίσω ορισμένα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για κατάρτιση, το, το, το, θέμα των διαφόρων σχόλων. Ε, ε, χωρών ε, και το κατά πόσον αν θέλετε οι τίτλοι σε επίπεδο αθλητισμού μπορούν να χρησιμεύσουν ιδιαίτερα. Μιλήσατε για την διπλή καριέρα και αυτούς τους αθλητές που όταν τελειώνει η καριέρα τους ως αθλητή μένουν ξεκρέμαστοι χωρίς τίποτα. Καταλαβαίνετε, μας απασχολεί πολύ το ζήτημα αυτό. Η κατάρτιση λοιπόν των αθλητών νομίζω ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Επίσης, όσον αφορά το ντόπινγκ. Ε, νομίζω ότι ορισμένες φορές ε, σκεφτόμαστε μόνο το ντόπιν ε, στους αθλητές υψηλού επίπεδου. Αλλά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με, με τα γυμνάσια, ε, με τους αθλητικούς συλλόγους, ε, τα γυμναστήρια κτλ. Τι μπορεί να γίνει εκεί με τους νέους. Και επίση, η διπλή νομοθεσία που υπάρχει πολλές φορές. Δηλαδή, όταν ένα αθλητής ε, βρεθεί να το πάρετε, ε, ε, υφίσταται κυρώσεις, αλλά βεβαίως επειδή σε επίπεδο αθλητικό, αλλά επειδή ο αθλητισμός δεν είναι υπεράνω του νόμου, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να ακολουθήσει και δίωξη ενώπιον δικαστηρίων. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα μερικές φορές. Αυτό θέλω να ρωτήσω και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, υπάρχουν κονδύλια για να προωθηθούν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες στο Βέλγιο. Έχετε αναλάβει δύο σημαντικές αρμοδιότητες και αυτό είναι πολύ καλό. Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε ποια θα είναι τα αποτελέσματα ε, ε, των, συνεδρίων, των διασκέψεων που θα οργανώσετε και όλων αυτών των συζητήσεων που έχετε προβλέψει και με πολύ ικανοποίηση άκουσα, σας άκουσα να λέτε ε, πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί μετά το τέλος της αθλητικής σταδιοδρομίας μια άλλη σταδιοδρομία για τους αθλητές Τι σκέφτεστε λοιπόν για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 3 εκατομμύρια ευρώ για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ελπίζω ότι θα το υποστηρίξετε και αυτό το πρόγραμμα. Θα είμαι σύντομος οι πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα που ανακοινώσατε είναι πάρα πολύ καλά, είναι σαφές ότι αγαπάτε τον αθλητισμό για, το, για την Ουάντα. Στη διάρκεια της ε, Προεδρία σας νομίζω ότι θα χρειαστεί να προωθήσετε αυτές τις σκέψεις ώστε να αναλάβει πιο ουσιαστικό μέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη Οάντα. και να υπάρχει ενδεχομένως και ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Οάντα. 50% των, χρηματο, χρημάτων, των κονδυλίων της Βουάντα παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συγκαλέσετε μία διάσκεψη υπουργών αθλητισμού, αν ναι, συνιστώ να καλέσετε και τους εκπροσώπους των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών διότι έτσι θα, έχει, θα συνδυάσετε ε, εκπροσώπους του, της διοίκησης του αθλητισμού και των ε, ομίλων και των ε, σωματείων. Τώρα το θέμα των στοιχημάτων. Ε, είναι παγκόσμιο φαινόμενο με αρνητικά στοιχεία γίνεται, υπάρχει μαύρη αγορά, υπάρχει, ε, υπάρχουν τα μονοπόλια που δημιουργούνται σε εθνικό επίπεδο, τα στημένα παιχνίδια, μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτόν τον τομέα, αυτή τη δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ θα ήμουν υπέρ. Τι πιστεύετε εσείς. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω, Υπουργέ, ότι στην αρχή ανησυχούσα λίγο, γιατί βλέποντας ε, ε, όλα αυτά τα μεγάλα επιχειρήματα, ε, χρηματοδότηση, προπολογισμό, εργασία, προγραμματισμό. Ε, ακούσαμε του προκάτοχου σα, του προραλήσοντε και φοβόμαι ότι ο αθλητισμό έρχεται σε τελευταία μοίρα. Ακούγοντά σα όμω βλέπω ότι πραγματικά το έχετε θέσει ω προτεραιότητα. Τώρα, επειδή οι άλλοι συνάδελφοι με κάλυψαν, δεν θα επαναλάβω αυτό το θέμα του ενό εκατομμυρίου του ευρώ και πώ θα κάνουμε όλα αυτά. Πώς θα καταφέρουμε λοιπόν. Και ε, είναι πολύ ε, ε, σημαντικό το θέμα αυτό και θα πρέπει να το δούμε. Τώρα, να ρωτήσω πολύ γρήγορα κάτι. Εσείς αναφε... κάνατε έτσι μια ανοίξη ε, για τον εθελοντισμό και τον αθλητισμό. 2011 θα είναι η Ευρωπαϊκή Χρονιά για τον εθελοντισμό. Επειδή φέτος λοιπόν έχουν ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το θέμα αυτό, ρωτώ, κατά την άποψή σας ε, υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια για συγκεκριμένα προγράμματα προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ah, right. I cannot see your name. Yeah. Α, δεν μπορούσα να διαβάσω το όνομά σας, γι' αυτό είχα ένα πρόβλημα. Σκροντεύσκα. Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Είναι δύσκολο πραγματικά να διαβάσετε το, να διαβάσετε το όνομά μου, το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που θίγει μια σειρά σημαντικών ε, θεμάτων. Αναφερθήκατε στην ε, συνάντηση των Υπουργών Αθλητισμού και ε, αναφερθήκατε διάφορες προτεραιότητες. Παραδείγματος την ιδέα του fair play και το θέμα του ντόπινγκ. Ε, δεν ξέρω ποια θα ήταν τα συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσε να αναλάβει εδώ η Βελική Προεδρία για να αντιμετωπίσει αυτά τα δύο προβλήματα. Αναφερθήκατε και στον εθελοντισμό. Έχετε κάτι συγκεκριμένο να προτείνετε. Αναφέρατε επίσης ότι θα πρέπει οι επόμενες προεδρίες να ακολουθήσουν στην ίδια άγουσα όπως εσείς. Και επίσης μέσα στις πρωτοβουλίες σας θα υπάρχει και η δυνατότητα να αναφερθείτε και στον αθλητισμό για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η είπατε ότι στη δήλωσή σας ότι ο αθλητισμός συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Εγώ έχω επισκεφθεί σχολεία και πανεπιστήμια και τους λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα για τα θέματα του αθλητισμού μιλάμε για τη, συζητάμε για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων. Για, αυτά, για αυτές χρειάζονται χρήματα, αλλά αυτές οι εγκαταστάσεις είναι σημαντικές διότι ε, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού. Χρειαζόμαστε όμως και ε, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας για τα νέα παιδιά. Τι πιστεύετε γι' αυτό. Είχα και κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά το ξέχασα. Σας ευχαριστώ. Λέω κύριο Σκέλη, δεν είχα ζητήσει το λόγο μέχρι στιγμή, αλλά άκουσα με μεγάλη προσοχή και πρέπει να σα πω ότι είχα κάποιε αμφιβολίε. Όχι απέναντι ε, στην Βελική Προεδρία, αλλά απέναντι σε κάθε Προεδρία, λαμβάνοντα υπόψη το, τη Δίκη τη Λισαβόνα και τα νέα εργαλεία και τα νέα μέσα και, το, και τις που θα έχουν όλα αυτά στη συνολικότερη, στην ευρύτερη εικόνα της στρατηγική 2020. Πρέπει να σας πω όπως ότι ε, ε, ε, αισθάνομαι αισιοδοξία μέσα από αυτά που άκουσα, γιατί υπάρχει ένα ρεαλιστικό στοιχείο. Πρώτα απ' όλα ε, μιλήσατε για ένταξη όλων αυτών στη στρατηγική 2020 και όσον αφορά την κάλυψη των κενών σε αυτά που ήδη ξεκινήσει, η διαδικασία της Μπολόνια, ε, πανεπιστήμια, ε, νεολαία σε κινητικότητα, όλα αυτά τα υποστηρίζω. Ο ε, όμως, μην ξεχνάμε ότι ε, ε είναι μια ευρύτερη εικόνα, γιατί εδώ πρόκειται για νέε αρμοδιότητε. Και εσεί μιλήσετε πραγματικά για ζητήματα τα οποία μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Προσωπικά, δεν θα ήθελα να σταθούμε πολύ και δεν θα ήθελα να ξοδέψουμε καθόλου χρήματα, αν θέλετε, στο θέμα του ντόπινγκ. Γιατί αυτό είναι ευθύνη τη ΓΟΑΝΤΑ. Και ενώ εμεί μπορούμε να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια αυτή, ε, είμαστε μια μικρή μειοψηφία εδώ. Εμεί θα πρέπει να βλέπουμε την ευρύτερη εικόνα και το πώ μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον αθλητισμό για να επιδράσει θετικά στι ζωέ των ανθρώπων. Μου αρέσουν ιδιαίτερα αυτά που είπατε, κυρίω το θέμα τη κοινωνική ενσωμάτωση μέσα του αθλητισμού, ε, τη ε, ε, κατάρτιση και τη προπόνηση, γυναίκε, ε, διαβίου, αθλητισμό, αθλητισμό για όλου. Άλλοι επίση αναφέρθηκαν στον αθλητισμό, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Και τέλο, βεβαίω, αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφό μου, κ. Λόκαρτ, κ. Σκούρια Πρέπει να ε, πραγματικά ε, ε, να ε, καταβάλουμε μια προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή ε, και το θέμα του προπολογισμού. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ κύριε Καλπές. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας παρόλο που θεωρώ ότι αναφερθήκατε κυρίως για ελιτιστικό αθλητισμό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα είναι η άλλη πλευρά, ο καθημερινός αθλητισμός, ο αθλητισμός των μαζών, γιατί εκ παραλλήλου προς τον πολιτισμό και ο αθλητισμός είναι ένα μέσο κατά της κοινωνικής, του κοινωνικού αποκλεισμού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνους που βρίσκονται περιθωριοποιημένοι στην κοινωνία είναι λοιπόν μια ευκαιρία για όλα τα παιδιά που μπορούν έτσι να ανοίξουν, να ενταχθούν στη κοινωνία μέσω του αθλητισμού. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω μέσα στα πλαίσια του, της γιατί η Ουγγαρική Προεδρία θα που θα σας ακολουθήσει έχει τις ίδιες απόψεις. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι το... οι δωρητέ ε, στον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιο μέσο ελέγχου που θα χρησιμεύει στην ε, εφαρμογή μιας δαφάνειας και υπέρ του αθλητισμού και υπέρ ονομιμών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, τελευταίος, εξίσου σημαντικός βέβαια, ο Ιβό. Eh, Ευχαριστώ, ε, Doris. Σε ένα λεπτό είπατε θα, θα μιλήσουμε. Ωραία. Θα προσπαθήσω να το κάνω. Έχουμε εδώ ένα νέο πρόγραμμα της Κομισιόν. Έχουμε τεράστιες, θα τεράστιες ευκαιρίες να παίξουν ένα ρόλο. Αναφερθήκατε σημασία του αθλητισμού στον, ε, στην κοινωνία. Είσαστε αθλητής κι εσείς και γι' αυτό θα μπορέσετε να ε, εργαστείτε επιτυχώς και προσβλέπουμε βέβαια και στην Ουγγρική Προεδρία συζητήσαμε για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και να τους βοηθήσουμε μέσα στο σωματεία τα αθλητικά, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αναφερθήκατε λοιπόν το θέμα του αθλητισμού και κοινωνία ε, και υπάρχουν όμως και αρνητικές επιπτώσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με τον κύριο Κέλλη ότι δεν είναι τόσο σημαντικό το ντόπι γιατί αφορά μόνο ένα μικρό ποσοστό των αθλητών. Είναι σημαντικό να καταπολεμηθεί γιατί βλάπτει την εικόνα του αθλητισμού σημαντικά. Είναι ενδιαφέρον αυτό που είπατε, να υπάρχει μια ευρωπαϊκή φωνή στην Ουάντα. Εντάξει, το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε και εμείς τι μπορούμε να συμβάλλουμε. Ε, κοιτάξτε όλους τους διάφορους ε, κανονισμούς που υπάρχουν στα 27 κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να ευθυγραμμιστούν και να υπάρχει σύγκληση των ε, νομοθεσιών. Υπάρχει η υπόθεση Μπερνάρ που παίζει εδώ ένα ρόλο. Και τέλος ο προπολογισμό. Κυρία Πακ, είπατε ότι δεν είναι φυσιολογικό να περικοπεί ο προπολογισμό. Τώρα που έχουμε περισσότερε αρμοδιότητε μέσα στα πλαίσια τη ε, συνθήκη τη Λισαβόνα, θα ήταν παράλογο να περικοπεί ο προπολογισμό. Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ναι. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Um, Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολλές ερωτήσεις, προσπάθησα να τις σημειώσω όλες. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Υποστηρίξατε το πρόγραμμά μας με τις παρεμβάσεις σας και θα ξεκινήσω με το θέμα του προϋπολογισμού. Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάμε για χρήματα, για δημοσιονομικά θέματα σε αυτή την ευαίσθητη δύσκολη περίοδο. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες σας. Τις αντιλαμβάνομαι απόλυτα και θα τις έχω κατά νου όταν θα συνομιλώ με τους ε, συναδέλφους μου. θα είναι δύσκολες οι συνεννοήσεις με τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. αναφερθήκατε στο ντόπινγκ, στον Ουάντα. Καταλαβαίνω τι λέει ο κύριος Κέλλη όταν ε, μου λέει ότι αυτός είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Δεν λέω ότι χρειάζεται διαφορετική συμφωνία. Δεν λέω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παράλληλο με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με τον Ουάντα αλλά πρέπει να δούμε ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας του Οάντα. Πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο εφαρμόζεται η συμφωνία αυτή με όσο γίνεται πιο ομοιόμορφο τρόπο. Έχει αποδώσει, ε, έχει δώσει καλά αποτελέσματα ήδη στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας και πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση ε, με τρόπο ενωμένοι με σαν ενιαίο μέτωπο. Δεν λέω να περάσουμε νέους κανονισμούς, νέους νόμους. Απλώς πρέπει να στηρίξουμε αυτά που έχουν ήδη αρχίσει και θα το κάνω αυτό σε στενή επαφή και διαβούλευση με τους συναδέλφους. Ε, τέθησαν ερωτήματα που αφορούσαν συγκεκριμένες δράσεις. Κάποιος μίλησε για ένα τουρνουά ποδοσφαίρου μεταξύ σχολείων. Πολύ ωραία ιδέα αυτή για να δούμε βεβαίως και τι είναι εφικτό, τι μπορεί να γίνει στην πράξη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα μαθαίνουμε ημένα από τους δε. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τα σχέδια δράσης τα οποία αναφέρθηκα. Η Ουγγρική Προεδρία θα ασχοληθεί και αυτή με το θέμα του κοινωνικού, της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το να μαθαίνουμε από τους άλλους, το να εφαρμόζουμε καλά παραδείγματα που έχουν εφαρμόσει άλλοι είναι πράγματα που δεν χρειάζονται πολλά χρήματα και προσβλέπω στις επαφές και στις συνομιλίες που θα έχουμε με τον Ούγγρους συναδέλφους στο μέλλον. Δεν μπορώ να σας δώσω απαντήσεις για όλα τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε. Θα υπάρξει μία εκδοχή στο 2012 και 2013 στα πλαίσια ενός νέου προγράμματος για τον αθλητισμό και θα, με πολλούς στόχους που, που θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο που θα κάνουμε, να εκπονήσουμε και να διαμορφώσουμε αυτό το, το πρόγραμμα αθλητισμού. Τα αθλητικά διπλώματα, τα αθλητικά πτυχία, ο κύριο Φίσας νομίζω αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Συμφωνώ με, αυτά, αυτό που είπατε. Και είναι καλή ιδέα. Αθλητικά πτυχία τα οποία θα αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο πρέπει να εστιάσουμε τις ε, προσπάθειές μας. Μετά το 2012 ε, ε, προβλέπεται ενδεχομένως να εφαρμόσει ένα προβλέπει δυνατότητα χρήσης αυτών των αθλητικών πτυχίων ανάμεσα στις διάφορες χώρες για το ντόπινγκ πολύ σοβαρό πρόβλημα Πρέπει λοιπόν να θέσουμε, να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Ελπίζω ότι αν οι νέοι βλέπουν τι συμβαίνει στην αγωνιστική και αν οι πρωταθλητές και οι κορυφαίοι αθλητές μπορούν να δώσουν το καλό παράδειγμα στα νέα παιδιά που ασχολούνται, αρχίζουν να ασχολούνται με τον αθλητισμό και αν τηρείται αυστηρά η συμφωνία του Βάντα είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε, θα πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Ήδη δεν υπάρχει, υπάρχουν αποκλήσεις ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη για το πώς εφαρμόζονται οι κανονισμοί της ΟΑΝΤΑ και θα καταβάλω προσπάθειες ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη εναρμόνιση σε αυτό το τομέα. Αθλητισμός και χρηματοδότηση μπορεί κανείς ε, και να έχει και αυτές τις δύο αρμοδιότητες. Κάποιος ρώτησε. Ναι, γιατί η εργασία και η απασχόληση και ο αθλητισμός είναι δύο τομείς οι οποίοι συνδέονται κατά κάποιο τρόπο μεταξύ τους εφόσον οι αθλητές πρέπει μετά από το, το αν τελειώσει η θεατρική σου διαδρομία να αναλάβουν κάποια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Και αυτή η διπλή κατάρτιση, η αθλητική και η επαγγελματική, χρειάζεται να, πρέπει να χρηματοδοτηθούν υπήρξε μια ερώτηση για το κατά πόσο θα έπρεπε να ενισχύσουμε την ε, προσώπησή μας στον ΟΑΝΤΑ. 25% της χρηματοδότησης προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το συζητήσουμε με τους συναδέλφους αυτό το Νοέμβριο, να υπάρξει μια ε, σημαντική ισχυρή δήλωση για αυτό το θέμα. Η Ισπανική Προεδρία τα πήγε πολύ καλά και ελπίζω ότι και εμείς θα μπορέσουμε να είμαστε σαφέστεροι στο μέλλον. Εάν υπάρχουν πέντε σε μία συνεδρίαση, το είδα το Μάιο στην τελευταία συνεδρίαση, μπορεί κανείς να καταφέρει περισσότερα αν παρίστανται ε, πολλά περισσότερα άτομα που προσπαθούν όλα να ακουστεί η φωνή τους. Είναι καλύτερο να υπάρχουν λίγα άτομα με ισχυρότερη φωνή. Στο Βέλγιο οι επιστήμες είναι κάτι που αντιμετωπίζεται σε ε, ομοσπονδιακό επίπεδο, ενώ ο αθλητισμός αντιμετωπίζεται σε περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε μια κοινοτική προοπτική, μια κοινοτική προσέγγιση Είπατε ότι το πρόγραμμά μας είναι φιλόδοξο, είναι πράγματι φιλόδοξο. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε, θα καταφέρουμε να πετύχουμε τα περισσότερα από αυτά που έχουμε προβλέψει, γιατί είναι σημαντικό να βάλουμε ψηλά το πύχη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και ελπίζω, ελπίζω πραγματικά ότι θα υλοποιήσουμε πολλά από αυτά που έχουμε κατά νου. Για τον εθελεντισμό δεν έχω τίποτε συγκεκριμένο να σας πω αυτή τη στιγμή Εν πάση περιπτώσει το έτος ε, του εθελοντισμού είναι το 2012. Με αυτό θα ασχοληθούμε λοιπόν αργότερα. Θα συναντηθούμε με την ε, Ουγγρική Προεδρία γιατί θα ε, αναλάβει τότε εκείνη την Προεδρία και θα συντονιστούμε με την Ουγγρική Προεδρία για να προωθήσουμε αυτό το θέμα του εθελοντισμού. Κάποιε υποδείξει θα μπορέσουμε να δώσουμε σε στενή συνεργασία, επαναλαμβάνω και πάλι, με την Ουγγρική Προεδρία, η οποία θα είναι κατεξοχήν αρμόδια για αυτό το θέμα. Εθλητισμός για όλους. Πάρα πολύ σημαντική δραστηριότητα, διότι συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική ενσωμάτωση όπω είπα είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα από τα σημαντικότερα ίσω στοιχεία. Δεν μιλάω μόνο για πρωταθλητισμό, μιλάω για το ερασιτεχνικό αθλητισμό που είναι που στον, στον οποίο αποδίδουμε την ίδια σημασία όπως και στον πρωταθλητισμό. Ελπίζω να το τόνισε αυτό επαρκώς στην ομιλία μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Εν αντιθέσει από κάποιον που το αμφισβήτησε, νομίζω ότι κάποιο που είναι υπουργό αθλητισμού και οικονομικό είναι ακριβώ ο σωστό. Γιατί μπορεί να πείσει τον Υπουργό Οικονομικών πρέπει να ταπανηθούν χρήματα για τον αθλητισμό. Για του άλλου είναι πιο δύσκολο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και σα ευχόμαστε για την εργασία σας κάθε επιτυχία. Είμαστε στο πλευρό σας, ιδίως όταν αφορά το θέμα την, ε, ε, την ενσωμάτωση ε, μέσω του ελθισμού και ακριβώς στην Νότιο Αφρική το είδαμε τελευταία ε, πώς ε, μπορούν τα παιδιά μέσω του αθλητισμού, μέσω του ποδοσφαίρου να πιστούν να συμμετάχουν και σε άλλους τομείς. Αυτό είναι πάλι πολύ χρήσιμο και ιδίως το ποδόσφαιρο. Και ακριβώς εδώ ε, μπορούν να εμπλακούν και παιδιά από ε, ε, οικογένειες μεταναστών. Σας ευχαριστώ λοιπόν και θα ξαναειδωθούμε σίγουρα κάποια στιγμή στο εξάμεινο και οπωσδήποτε στο τέλος, όταν θα μπορέσουμε να σας συγχαρούμε. Κάθε επιτυχία. So, jetzt schließen wir diese Sitzung und ich darf die Koordinatoren bitten, hier zu sein. Morgen früh um 9 sind alle wieder eingeladen. Λοιπόν, κλείσει την τρεις εδώ, συντονιστές μετά. Κύριε Φάρα, παρακαλώ. Sie möchte gerne das verschieben, muss ich offiziell.